Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ε, ας ξεκινήσουμε. Καλώς ορίσατε. Πρώτα απ' όλα, ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εδώ υπάρχει μία μικρή αλλαγή όσον αφορά το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Ο αντιπρόεδρος μας, ο κ. Δασεβόσκη, ο εισηγητής, ε, και οι δύο ε, σκιώδεις θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επεξεργαστούν τους, ε, τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά το 10, την έκθεση Βοσεβόσκη, την αναβάλουμε για τις 18-19 Δεκεμβρίου. Αν δεν έχετε λοιπόν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη με αυτή την ε, τροποποίηση. Κατά τα άλλα, θέλω να ενημερώσω τους συντονιστές ότι αν σήμερα κατορθώσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, στο τέλος της σημερινή συνεδρίασης θα συνεδριάσουν τονιστές, αντί για αύριο δηλαδή που προβλέπετε. Και έτσι θα κερδίσουμε χρόνο γιατί αύριο θα είναι πιο πιεσμένη η ημέρα μας. Επίσης ε, θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής. Σημείο υπαριθμών 2. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά και για την συνεδρίαση 14η Μαΐου και για τη συνεδρίαση της 30η-31η Μαου. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι η σημερινή συνεδρίαση ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ε, παρουσιαστεί ήδη 610 τροπολογίες ε, σχετικά με το φάκελο για τις άμεσες πληρωμές και 140 τροπολογίες για τον κανονισμό σχετικά με την ε, ενιαία, ε, την κοινή αγορά. Φτάνουμε δηλαδή γύρω στις χίλιες, ε, γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε να περιορίσουμε λιγάκι τον αριθμό των τροπολογιών. Και επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία θέλω να σας υπενθυμίσω ε, το σημείο της γραμματείας όσον αφορά τον τρόπο ε, παρουσίασης ε, τροπολογιών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κατά τα άλλα, Είμαι ευτυχής που μπορώ σήμερα να δεχτώ, να δεχτούμε στην Επιτροπή μας μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από τη Νέα Ζηλανδία της οποίας προείσταται ο κύριος Λόκουτ Σμιτ πρόεδρος της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά αγαπητοί φίλοι από τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω και την ε, ομάδα επισκεπτών από την Τοσκάνη, από την Ιταλία. Καλώς ορίσατε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης, ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις ε, για το μελλοντικό για το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι καθοριστική σημασία για την κοινή γεωργική πολιτική και για τις προτάσεις ε, μεταρρύθμισης τις οποίες και εξετάζουμε. Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω ότι πριν από 10 ημέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε ε, συζήτηση για το περίφημο Negotiation Box το οποίο παρουσίασε η Δανική Προεδρία. Στα συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής δεν αναφέρονται ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία για το πολιτές δημοσιονομικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δική μας άποψη, αυτή που θα ακούσουμε σήμερα και την οποία και θα συζητήσουμε, η άποψή μας λοιπόν είναι κατ' ουσίαν μια ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την ε, βούληση της δικής μας Επιτροπής ε, που εκφράζουμε ε, προς την Επιτροπή Προλογισμών σχετικά με τα στοιχεία που υπάρχουν. Επιθυμούμε δηλαδή τα στοιχεία αυτά να συμπεριληφθούν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε μία ευκαιρία για να επαναλάβουμε και επιβεβαιώσουμε τη βούληση του Κοινοβουλίου. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι σημείο κίνησης είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εκφράστηκε στα ψηφίσματα της 8ης Ιουνίου του 2011. Πρόκειται για την περίφημη έκθεση Σούρε και τις 23 ε, Ιουνίου του 2011 πρόκειται τη δική μας έκθεση Albert Dess. Και στις δύο λοιπόν αυτές τις ε, περιπτώσεις και στην Επιτροπή Σούρε και στη δική μας την ε, έκθεση Dess το, το Κοινοβούλιο ζήτησε με απόλυτη σαφήνεια ο ισολογισμός της κοινή γεωρικής πολιτικής να παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο που είναι σήμερα και σε ε, πραγματικούς ε, αριθμούς. Έτσι λοιπόν η δική μας άποψη παραμένει η ίδια. Αυτή είναι η θέση μας. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν. Νομίζω ότι είδα τον διευθυντή κύριο Μέγγελ. Και σας υπενθυμίζω ότι αν υπάρχουν τροπολογίες για αυτή την γνωμοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Ε, βλέπω ε, τον κύριο Λαμπία, κοιτάξτε, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα. Και η ε, γνωμοδότηση αυτή, όπως σας είπα, θα υπογραμμίσει απλά την απαρασάλευτη βούλησή μας. Θα ήθελα να πω στους αδέλφους, αν θέλουν να λάβουν το λόγο πρέπει να το δηλώσουν. Ντελάνς και Λαβία έχουν ήδη δει το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή κύριο Μόγγελ. Η Έστερ είναι η πρώτη που θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έγγραφα εργασία που μας στείλατε και στο οποίο γίνεται μια παραπομπή της στην έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Εγώ είμαι εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ και Είπατε ότι αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλεί ως πάγωμα του προϋπολογισμού ανταποκρίνεται στην ουσία, αντιστοιχεί στην ουσία σε μία μείωση 10%. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή αυτού του ε, μειωμένου προϋπολογισμού στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης ε, να σκεφτούμε και μια θέση αναδίπλωσης. Φυσικά, ε, μένουμε στην έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε και την πραγματικότητα. Γιατί θα ληφθούν και αποφάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ ταυτόχρονα η κρίση σοβεί. Και η θέση των κρατών μελών είναι σχετικά ασθενής και η προβολή της. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και τη συγχρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα. Αν τα κράτη-μέλη δεν διαθέτουν αρκετά κονδύλια για να συνεισφέρουν στον κοινοτικό προπολογισμό, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη να προσθέσουν κάποια κονδύλια. Σε ό,τι αφορά το ΕΛΚ, για το δεύτερο πυλώνα ήδη προβλέπουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις για να μην περικοπεί αισθητά ο προπολογισμό για τη γεωργία. Επίσης, ίσως θα πρέπει να προσελκύσουμε το συντομότερο δυνατό ιδιωτικά κονδύλια, ιδιωτική χρηματοδότηση, ένα μέσο που ελάχιστα το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει σε αδρές γραμμές στο κείμενό σας, αλλά θα μπορούσαμε να το συμπληρώσουμε και να δούμε και τη γραμμή αναδίπλωσή μα. Πολύ ωραία, Έστερ. Και ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά σου τα σχόλια και είναι σαφές ε, ότι θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτά τα στοιχεία. Ο Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να πω κάτι έτσι πιο ευρύ όσον αφορά το κείμενο της έκθεσης. Πρόκειται για τις ε, νέες ε, δημοσιονομικές ε, προοπτικές γιατί νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας δεν νομίζω ότι προχωρήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Και από την άλλη θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε βήματα προς τα μπρος υπό την Κυπριακή Προεδρία. Σήμερα το πρωί συμμετείχα σε μία τριμερή συνάντηση για τον προπολογισμό του 2013 και αποκόμισα την εξής αίσθηση, ότι βρισκόμουν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Διότι αν από τη μία πλευρά στις 28 και στις 29 το Συμβούλιο μίλαγε για κατευθυντήριες γραμμές στην ανάπτυξη και την απασχόληση, από την άλλη το Συμβούλιο περιέκοψε ε, κατά 17% τη, τα κονδύλια για την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη. Άρα δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν γνωρίζει δεξιά τι πει αριστερά. Κατά τα άλλα, ε, αυτή την εμπειρία έκανα σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, μακριά και πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα. Διότι από τη μία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, βλέπω ότι έχουμε έναν τεράστιο όγκο ε, τροπολογιών για την έκθεση Επιτροπής και για την έκθεση των συναδέλφων, τις εκθέσεις των συναδέλφων. Από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν προχωράει γρήγορα. Και μόνο αυτό, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μια σημαντική καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων σε σχέση με αυτά που είχαν προβλεφτεί πριν από κάποιες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν φτάνω στην εξή σκέψη. Ίσως θα έπρεπε με την Επιτροπή να αξιολογήσουμε τι θα έπρεπε να κάνουμε, το σενάριο δηλαδή, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια εναλλακτική λύση για την κοινή γεωργική πολιτική. Διότι ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις, ενδεχομένως να υπάρξει κάποια σύγκρουση ανάμεσα στα τρία όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με αυτό που σας είπα, Πρόεδρος από ό,τι φαίνεται ε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θετικές ε, ευχάριστα νέα και ίσως αυτό να ισχύει και για το Eurogroup που θα συνέλθει σήμερα. Πάντως το Κοινοβούλιο θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει χρόνο. Όμως θέλω να πω ότι αν δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την κοινή γεωργική πολιτική δεν θα είναι και εύκολο να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος George Lyon. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έγγραφο όσον αφορά την Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης. Γιατί αν δούμε τι έχει να πει η ομάδα εργασίας και η ομάδα επαφής όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συντοποιούμε ότι οι απόψει είναι ξεκάθαρες. Οι συμβιβασμοί θα πρέπει να ψηφιστούν και στη συνέχεια δεν θα περάσουμε στην ε, Ολομέλεια ή δεν θα φτάσουμε στην Ολομέλεια με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα. Πρέπει λοιπόν εμείς να καταφέρουμε να εκφράσουμε σαφώς την απόψή μας πού θα βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές όσον αφορά σημαντικά δημοσιονομικά ζητήματα. Πρέπει ξεκάθαρα να εκφράσουμε την άποψή μας στην γνωμοδότηση αυτή, γιατί διαφορετικά οι διαπραγματευτές οι οποίοι θα ευασιστούν στην έκθεση ΣΟΥΡ ως βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το περιεχόμενο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και τον σχετικό συμβασμό, δεν θα καταφέρουν να καλύψουν όλα τα ζητήματα τα οποία εμεί θέλουμε να καλύψουμε. Δεν καλύπτονται όλα στην έκθεση ΣΟΥΡΕ, όλα τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Επομένω, θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να διευθετήσουμε καλύτερα τα πράγματα και να εκφράσουμε την θέση μα. Όσον αφορά το προπολογισμό, έχουμε επίση μια πολύ καλή ευκαιρία για να πούμε πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές. Συντοπιώ ότι ε, θέλετε να διατηρήσετε το προπολογισμό σε προηγούμενα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι έχουν γίνει σημαντικές περικοπές ε, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν πρέπει να βρεθούν ακόμα περισσότερες εξοικονομήσεις, τότε τουλάχιστον αυτές δεν θα πρέπει να προέλθουν από την κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του πολιτού πλαισίου. Πρώτον αυτόν, Δεύτερον, δεν ξέρω αν θα πρέπει να συζητήσουμε για το ζήτημα της κατανομής. Πάλι η έκθεση Σούρε δεν αναφέρεται καθόλου στο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν εμείς θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια γενικότερη θέση χωρίς να επισέλθουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο συνάδελφος Κάπουλας Σάντος. Μου δίνεται πάντω η εντύπωση ότι και από αυτού θα πρέπει να πούμε κάτι, να δούμε δηλαδή, να πούμε ποια είναι η απόψή μα όσον αφορά το ζήτημα τη επανακατανομή. Τρίτον, τα όσα βρίσκονται εκτό πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου και τα όσα βρίσκονται εντό του πλαισίου αυτού. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση και τη ψηφορία ακόμα, δεν ελήφθησαν υπόψη κάποια κονδύλια όσον αφορά το EGF ή όσον αφορά έκτακτες περιστάσεις. Θεωρείτε ότι είναι αυτή η σωστή προσέγγιση ή μήπως ε, η Επιτροπή μας θα επιθυμούσε τελικά να καλύψει με την άποψή της, με την γνωμοδότησή της όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία στην ουσία υφίστανται. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν, να επανέλθουν, να επιστρέψουν στον προπολογισμό. γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ενταχθούν και πάλι στον προπολογισμό, δεν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά κονδύλια, τότε ουσιαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάλι μία περίπτωση περικοπής ε, κονδυλίων. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να πούμε ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ, ποια είναι η βάση διαπραγμάτευση για μα ω Επιτροπή Γεωργία και Ανάπτυξη τη Υπαίθρου. Σα ευχαριστώ πάντω για την γνωμοδότησή σα και με το αρχικό σα έγγραφο θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση συζήτηση. Πρέπει απλώ τώρα στη συνέχεια να δούμε ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αν υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει και θα ενταχθούν στη συζήτηση. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σα. Η μόνη λοιπόν δυνατότητα που έχουμε για να προβάλλουμε την άποψή μα σχετικά με το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αυτό που είπατε εσεί. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση γιατί βλέπω ότι έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι ο κύριος Κάπουλα Σάντο και μετά ο κύριο Μαγκίνε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εγώ απλώς θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους εγκομίασαν το έργο σας και νομίζω ότι το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Λάιον είναι πολύ εύστοχο. Το έγγραφο της Δανικής Προεδρίας κάνει λόγο για την ε, ανακατανομή. Και είχαμε μια πρώτη θέση των ε, Υπουργών για το θέμα αυτό. Οπότε θα συμπλήρωνε το έγγραφο αυτό το ζήτημα που είναι από τα πιο ε, ευαίσθητα από πολιτική άποψη για το οποίο θα πρέπει να συσπυρώσουμε τις προσπάθειές μας για να το διαθετήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρω τις ανησυχίες μας και τη συζήτηση στην Επιτροπή. Γι' αυτό και σας συγχαίρω για το έργο σας, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Συνάδελφοι, πρέπει να ε, πω κάτι ότι τώρα ήρθαν οι Νεοζηλανδοί. Όταν τους ε, καλωσορίσαμε και τους ε, χαιρετήσαμε, δεν ήταν ακόμα εδώ, γι' αυτό επανέρχομαι. Ε, καλωσορίζω λοιπόν τον συνάδελφο κ. Λόχουτ Σμιτ, που είναι ο πρόεδρος της Βουλής Αντιπροσώπων της Νέα Ζηλανδίας και καλωσορίζω όλους όσοι ήρθαν σήμερα εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Μάριο. Με τη Μάριο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και για το έγγραφο εργασίας. Δεν ξέρω θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και τους αδέλφους από τη Νέα Ζηλανδία αν είχαν ποτέ προβλήματα με τον προπολογισμό και τη γεωργία, με τη γεωργία μάλλον. Να πω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή για μένα. Είπατε ότι έχουν υποβληθεί περίπου χίλιες τροπολογίες. Θεωρώ ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Όλες αυτές οι τροπολογίες ζητάνε από τους αγρότες, ιδίω στα πλαίσια των άμεσων πληρωμών, να κάνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερη υποστήριξη. Η δική μου κόκκινη γραμμή είναι ακόλουθη. Αν ο προπολογισμό δεν μείνει εκεί πέρα που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, τότε ουσιαστικά θα μειώσουμε τις τροπολογίες αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ζητάμε από τους αγρότες να κάνουν περισσότερα πράγματα, να πιέσουν περισσότερο με το ζήτημα του πρασινίσματος και να τους δίνουμε και λιγότερα χρήματα παράλληλα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε. Ευχαριστούμε Μάριον, ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κοίταξε, εμεί ε, ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία και την έκθεση Αλμπερντές και την έκθεση της Επιτροπής Σούρε. Άρα δηλαδή αυτή η κόκκινη γραμμή πρέπει να μας ενώσει όλους. Η Μπρίτα Ρέμερς, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για το, το πραγματικά πολύ καλά δομημένο έγγραφο το οποίο ε, στοχεύει σε ορισμένα θέματα. Και θέλω να πω ότι εγώ φοβάμαι ότι μερικές φορές ε, η όλη αυτή η συζήτηση για την κρίση που γίνεται δεν ε, αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα ποσά τα οποία ε, κινούνται δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με το δικό μας τον προπολογισμό που είναι πάρα πολύ μικρός. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αγωνιστούμε περισσότερο για τον γεωργικό προπολογισμό. Γιατί αν θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερα στην Ευρώπη τότε τα ίδια τα κράτη-μέλη καταρχήν θα πρέπει να δείξουν ότι είναι επιθαρχημένα. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν πράττουν. Ω εκ τούτου λοιπόν χαίρομαι γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και στο τέλο ε, φαντάζομαι θα καταλήξουμε σε μια γραμμή την οποία θα στηρίξουν όλοι. Πολύ ωραία. Μπρίτα Ελίζαμπετ Κόσιγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά ε, που είπε η προλαλήσασα ε, σχετικά με τις ε, περικοπές του γεωργικού προϋπολογισμού. Ο κ. Ντελάγκε το είπε ότι ο τομέας της γεωργικής ανάπτυξης δέχεται τεράστιες πιέσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Οι Υπουργοί Οικονομικών θεωρούν ότι σε αυτόν τον προϋπολογισμό μπορούν να κόψουν πάρα πολλά κονδύλια. Ε, και εμείς ε, θα πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε ότι τα κονδύλια για την γεωργική ανάπτυξη είναι ε, αναπτυξιακά κονδύλια, πράσινα κονδύλια και επουδενή δεν θα πρέπει σε μια εποχή όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στον προπολισμό επουδενή δεν πρέπει να ενδώσουμε. Συμφωνώ ε, με την κυρία Μακίνες ε, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα και τις ε, άμεσες πληρωμές. Νομίζω ότι ο γεωργικός τομέας αξίζει περισσότερα και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ο Τζοβάνι Λαβία το είπε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστούμε και ένα εναλλακτικό σενάριο ε, για το τι ε, θα μπορούσε να συμβεί αν δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαπραγματεύσεις. Γιατί στις ε, άμεσες πληρωμές υπάρχει πρόβλημα. Ίσως ε, θα μπορούσαμε, αν χρειαστεί, να προχωρήσουμε με 12 αρτημόρια. Αλλά οι εξελίξεις... είναι πολύ σημαντικές για τους γεωργούς οι οποίοι αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια. Τα χαιρόμουν λοιπόν πάρα πολύ αν από πλευρά ε, Επιτροπή και από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγαμε σε συγκεκριμένε απόψει. Και κάτι που αφορά του ε, αριθμού. Πριν από λίγε μόνο εβδομάδε ε, δημοσιεύτηκε μία μελέτη η οποία ασχολείται με τις ε, γεωργικές πληρωμές ε, σε διάφορα κράτη του κόσμου. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλουν τριπλάσιες επιδοτήσεις ε, σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου, κυρίως να το επισημάνουμε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Το θέμα δεν είναι να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας ε, και την παραγωγή τροφίμων μόνο, αλλά να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που επουδενεί. δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρόεδρος, ε, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγνιού. Ε, Ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κύριο Λαβία, που δεν έχει το καθόλου αξιοζήλευτο έργο να βάλει κάποια τάξη και να βγάλει κάποιο νόημα από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Όπω είπε λοιπόν και ο κύριο Λαβία, παρά την άοκνη προσπάθειά του, και τον πιστεύω, είναι, είπε ότι αισθάνεται σαν να βρίσκεται σε αυτοκίνητο Χωρί οδηγό και το οποίο κατευθύνεται χωρί κανένα έλεγχο. Ο Winston Churchill θα έλεγε κάτι παρόμοιο, ότι είναι μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λαβία. Επίσης, ε, είναι ενισχυτική και η στάση της Δανία, γιατί είχε το πρώτο εξάμεινο του έτους, που ε, είχε ένα πλήρε εξάμεινο τη Προεδρία και πήγε ε, τελικά το. Η Δανία είναι γνωστή για την ε, γεωργία της, για την κτηνοτροφία τη, τη χειροτροφία ιδιαίτερα και τη γεωργία με το κρυθάρι, αλλά η Κύπρος έχει την πιο μικρή ε, το μικρό εξάμεινο, ε, γιατί μεσολαβούν οι καλοκαιρινέ διακοπέ, οπότε θα είναι κουτσουρεμένη ουσιαστικά η Κυπριακή Προεδρία. Άλλωστε, είναι μια χώρα που δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία με τη Γεωργία. Και παρόλα αυτά, αυτή θα διεκπαιρέσει το θέμα. Οπότε, ε, συμμερίζομαι την απορία του κυρίου Λαβία. Τι θα γίνει, ο χρόνο περνάει. Και ερώτηση προ την Ευρική Επιτροπή. Μήπω τελικά θα βρεθούμε και πάλι πρωτοτελεσμένο γεγονότα και θα μα επιβληθεί εκ των άνω μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ε, τα θέματα που αναφέρθηκαν είναι τα σημαντικότερα για τη δική μου την πολιτική ομάδα. Αυτά που είπε ο κύριος Τζοβάν Λαβία αλλά και άλλοι καταδεικνύουν ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνούμε και το είπε και η Μάριον Μαγκίνες ε, ότι ο ο γεωργικός ε, προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει σε ίδιο επίπεδο. Οι προτάσεις όμως της ε, ε, Κομισιόν σημαίνουν σημαντικές περιεκοπές. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός, το περίφημο αυτό 7% που συνεπάγεται μεγαλύτερες δαπάνες. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ για το ότι τα κράτη-μέλη μόλις ε, την τελευταία στιγμή δραστηριοποιούνται. Είμαι ε, βουλευτή σε 20 χρόνια και στις διαπραγματεύσεις ε, πάντα μας έλεγαν η συμφωνία επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή στο παραπέντε. Αν τα πράγματα τώρα αλλάξουν θα χαρώ πάρα πολύ αλλά δεν έχω και πολλές ελπίδες. Ενδέχεται την επόμενη χρονιά να υπάρξει κάποια αλλαγή ε, αλλά αυτό όμως θα είναι πολύ αργά. Δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί μεταρρύθμιση την 1η 1 η του 2014. Ε, αυτό η Κομισιόν ε, πρέπει να το έχει κατά νου και η γεωργική μεταρρύθμιση θα μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον έχει ξεκαθαριστεί και το θέμα της ε, χρηματοδότησης. Γιατί το να υπάρχει μεταρρύθμιση με 20% λιγότερους ε, πόρους, αυστηρότερους όρους και μεγαλύτερη γραφειοκρατία, εμείς αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Εμείς επιθυμούμε η γεωργία στο μέλλον να στηριχτεί όπως της αξίζει και αυτό δεν θα είναι μόνο υποστήριξη της ε, γεωργίας, ε, θα είναι ε, και ένα όφελος που θα προσποριστούν οι καταναλωτές. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι καταναλωτές θα έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θα αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων. Έτσι λοιπόν το να χρησιμοποιείτε αυτό το 1%. Αυτό είναι το ελάχιστο και πρέπει να σκίσουμε πίεση στα κρατημέλη έτσι ώστε να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Τώρα, επόμενος ομιλητής, ε, Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο από τα κράτη-μέλη ε, να μας ε, προτείνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις αλλά δεν αναφέρουν αριθμούς. Ε, αυτό δεν είναι σωστό. Το fair play λέει ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει τα κονδύλια. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι γίνεται συνεχώς λόγος για ανάπτυξη και απασχόληση. Και εγώ συμφωνώ αλλά όμως τη γεωργική πολιτική ε, την εξαιρούν όλοι. Και εμείς στον πρώτο πυλώνα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να συζητάμε για ανάπτυξη και απασχόληση. 17 εκατομμύρια ε, εργαζόμενοι στη γεωργία δεν είναι όμως αμεληταίοι. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρξουν νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και να παραμείνουν αυτοί που έχουν τώρα κάποια θέση. Η ε, κοινή γεωργική πολιτική λαμβάνεται σοβαρά υπόψη μόνο όταν επιδεικνύει συνέπεια και αυτό το έχουμε κατανοήσει. Κατά τα άλλα, για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν τελικά ο προϋπολογισμός ε, διαφοροποιείται σημαντικά από τις αρχικές μας ε, προτάσεις, τότε θα πρέπει και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι δυνατό το είπε ο συνάδελφος, να έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία και ε, λιγότερα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά παρακαλώ να παραμείνουμε συνεπείς, να είμαστε σκληροί στις διαπραγματεύσεις αλλά και τίμιοι όσον αφορά τη σχέση μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Μισελ Νταντέν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εργασία που κάνατε εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό. Το ζήτημα του προπολογισμού, καθώς επίσης και του προπολογισμού για τη Γεωργία, είναι κάτι που τελικά θα αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Γιατί το γεωργικό ζήτημα σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες προσπαθούν να συνδέσουν την εξισορρόπηση των γεωργικών επιδοτήσεων με τον γενικό συμβασμό που πρέπει να επιτευχθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε προς τις χώρες ακριβώς τι συμβαίνει, τι διακυβεύεται και ως προς αυτό θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή τη στιγμή προσπαθούμε από το 2002 να ακολουθούμε με ένα κοινό τρόπο. Το 2002 ήταν η τελευταία ημερομηνία που φασίσαμε για ένα κοινό προπολογισμό και θέλουμε ουσιαστικά να διατηρήσουμε ένα προπολογισμό για 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα προπολογισμό που είχε αποφασιστεί όμως για 15 χώρες μέλη. Την εποχή εκείνη θεωρούσαμε ότι η αγορά από μόνη της θα μπορούσε να επιλύσει τα γεωργικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν τροποποιηθεί. Βρισκόμαστε πλέον στον 21ο αιώνα, σε διαφορετικό κόσμο. Βλέπουμε ότι οι αγορές από μόνες τους δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις κρίσεις που έχουν δημιουργηθεί από την αυξομοίωση των γεωργικών τιμών. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν χώρες που στο παρελθόν ζητούσαν μείωση του γεωργικού προπολογισμού και τώρα είναι οι ίδιες οι χώρες αυτές οι οποίες δίνουν επιπλέον επιδοτήσεις στο γεωργικό τους κλάδο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη Βραζιλία, στην Αργεντινή αλλά θα μπορούσα να αφαιρθώ και η Ελιζαμπέθ Κεσιγκέρ το είπε, και στο τι συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στο παρελθόν μα ζητούσαν να κάνουμε περικοπέ και αν δούμε τα αριθμητικά του στοιχεία, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δίνουν περισσότερα κονδύλια, σίγουρα τα τριπλάσια ποσά. Νομίζω λοιπόν ότι απέναντι στην πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να βασιστούμε. Αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει να υπερασπιστούμε και ουσιαστικά δεν λέω να μην εξελιχθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Σαφώ θα πρέπει να εξελιχθεί και να τροποποιηθεί. Κάθε φορά που μιλάμε όμω για τα χρηματοδοτικά μέσα, θα πρέπει να έχουμε συγκρίσιμε καταστάσει και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο κόσμο έχει αλλάξει από το 2002. Δεν μπορούμε πλέον να αποτελούμε εμεί τα καλά παιδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα δεχόμαστε αγόγγιστα τα όσα μα ζητούνται, θα πρέπει οι αποφάσει μα να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και να λειτουργήσουμε συνειδητά και υπεύθυνα αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσει να επιτελεί τον σημαντικό της ρόλο η γεωργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, και εμεί ε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κατορθώσουμε, να διατηρήσουμε αυτή την κόκκινη γραμμή. Αντιπρόεδρος Σεκηγεύσκη. bardzo przepraszam. Ευχαριστώ. Φυσικά μεταξύ μας επικρατεί μεγάλη ομόνοια και συμφωνία γιατί ε, είμαστε συνδεδεμένοι με τη γεωργία, έχουμε ευαισθησίες για τη γεωργία, οπότε ε, υπάρχει σχετικά ομοφωνία μεταξύ μας. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαμορφώσουμε με ιδιαίτερο τρόπο την θέση της Επιτροπής γεωργία απέναντι στο προϋπολογισμό και απέναντι στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, γιατί η μεταρρύθμιση ΚΑΠ εντάσσεται και στις ε, νέε δημοσιονομικές προοπτικέ. Και μάλιστα ανακύπτει το ζήτημα. Τι θα κάνουμε πριν τι θερινέ διακοπές και τι μετά από αυτέ. Δεύτερο πρόβλημα, το διαπίστωσα αυτό και μεταξύ των Πολωνών Ευρωβουλευτών, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει και μεγάλη ε, γνώση για την ε, γεωργική πολιτική. Δεν γνωρίζουν όλοι οι ευρωβουλευτές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωργικής πολιτικής. Μια κάποια στιγμή έσβησε το μικρόφωνο του κυρίου Σεκέρσκη. Δεν υπάρχει λοιπόν γνώση σε όλους τους ευρωβουλευτές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Και επίσης ιδιαίτερα στο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε επίπεδο Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και εκεί έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις για τη Γεωργία. Από πού προέκυψαν όμως εκεί οι κατευθυντήρες γραμμές και ποιες ήταν η ε, προσεγγίση και των διαφορών χωρών και σε τι φάση τη βρίσκεται η διαδικασία, βρίσκεται σε προχωρημένη φάση. Είναι σημαντικό επίσης, ε, γιατί και επίσης, το θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εκεί αναφέρθηκαν θέματα είναι σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η θέση που θα θετήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Ε, εγώ, όπως είπε και ο κύριος ε, Νταντέν, ε, θεωρώ ότι δεν αναπτύσσουμε ιδιαίτερα μετά την διεύρυνση των προϋπολογισμών και αντί να, παρόλο τη διεύρυνση που είχαμε αντί να αυξάνεται ο προπολογισμό, φαίνεται ότι όλο και συρρυκνώνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σεκέρσκι, ο Ζωζέ Μποβέ και ο τελευταίος κύριο ε, κύριος Μάρτιν Χόισλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ θα κάνω μια παρέμβαση επί της ουσίας όχι προς την ίδια κατεύθυνση του Μισελ Δαντέν, μάλλον όχι με, τον, όχι με τον ίδιο τρόπο, ε, με τον Μισελ Ταντέν, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, συμφωνώ με τα επιχειρήματα των συναδέλφων, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους. Εμένα περισσότερα με ανησυχεί το θέμα τη νομιμοποίηση τη γεωργικής μα πολιτική. Αν η, γεωργική μα πολιτική δεν έχει νομιμοποίηση σε σχέση με τι προκλήσει που καλούμαστε να αποφάσεις, που, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, η κοινή γνώμη θα πει προ τι να συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε μια γεωργία που καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τι θέσει απασχόληση και δεν παράγει και ποιοτικά προϊόντα. Δυστυχώ, αυτό θα το μάθουν οι, οι Ευρωπαίοι πολίτε, γιατί πια έχουν δημοσιευθεί οι προτάσει. Και μάλιστα οι προτάσει ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δημόσιε. Και μάλιστα σήμερα αυτέ οι θέσει ε, πάνε σε λάθος κατεύθυνση. Και όταν βλέπουμε ότι δεν έχει προχαρήσει με ταχύ ρυθμό η κατανομή μεταξύ των χωρών και τα ανώτατα όρια που προτείνονται σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη κατανομής των ενισχύσεων ε, στη γεωρία και μάλιστα είναι μια προσβολή ιδιαίτερα για τους μικροκαλλιεργητές και αν δούμε τι συμβαίνει με το πρασίνισμα που αρχίζουμε και ξυλώνουμε το ένα μέτρο μετά το άλλο ε, Πώς θα πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι θέλουμε κονδύλια για μια γεωργία που στριμώχνει ε, τους γεωργούς συνέχεια και δεν συνάδει και με την αναβάθμιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να δώσω τώρα το λόγο στον Μάρτιν Όσλιν και μετά Μάνου Μακίνης ξαναζήτησε λόγο. Μάρτιν, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το θέμα έχει στηθεί επανειλημμένα, αλλά βέβαια εμένα ε, μου δημιουργεί πάντα εντύπωση. Εδώ οι συνάδελφοι είπαν ότι ανήκουν στην πολιτική οικογένεια των χριστιανοδημοκρατών και ίσως θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να παρουσιαστούν στο Βερολίνο. Διότι ειδικά η γερμανική κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία ασκεί τεράστια πίεση στον προπολογισμό των κρατών μελών. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον εδώ οι συνάδελφοι που έχουν ε, ε, κόμματα που κυβερνούν να τους πούνε ότι κοιτάξτε δεν γίνεται ε, αυτό το 1% να περικοπεί. Δεν είναι δυνατόν να ε, υπάρξουν περικοπές στον τομέα της ε, γεωργίας. Επίσης, η σχέση ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις και τα χρήματα εδώ και είναι σημαντική, γιατί αν δεν υπάρξει έγκριση μεταρρύθμισης, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο στο Κοινοβούλιο να υπάρχει έγκριση για τον συνολικό προϋπολογισμό. Δεν νομίζω ότι οι γεωργικές ε, ε, δαπάνες ε, θα παραμείνουν ως έχουν. Όλοι θα αντιμετωπίσουμε τεράστια πίεση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας κάνω απευθύνω έκκληση σχετικά με την μεταρρύθμιση να μην αναφέρετε ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό είναι ένα καθοδικό σπυροειδές και δεν πρέπει να το τροφοδοτούμε εμείς. Γιατί σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να κερδίσουμε σε αυτό το καθοδικό σπυροειδές των επιδοτήσεων προφανώ, καθοδικό, προφανώς προς τα κάτω. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να έχουμε αρκετά επαρκή κοντήλια. Ευχαριστούμε. Η Μάριον έχει δει το λόγο ξανά και τη στον δίνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που δευτερολογώ. Πάντως πρέπει να απαντήσω στα σχόλια του κυρίου Μποβέ. Προσπαθούσα να βρω αυτή τη στιγμή την μελέτη την οποία μας έστειλε για την άποψη της κοινή γνώμης όσον αφορά τη γεωργία. Ε, θέλω να πω ότι η άποψη κοινή γνώμης είναι ιδιαίτερα θετική. Και όταν μιλάμε για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, Διαφωνώ για πάρα πολλά πράγματα τα οποία είπατε για τη βιωσιμότητα, αλλά το να λέτε επίση ότι ο Ευρωπαίος πολίτη έχει αρνητική γνώμη για τη γεωργία, αυτό δεν στέκει, δεν αληθεύει και βασίζομαι στη μελέτη που μας στείλατε. Το ζήτημα της νομιμοποίησης τώρα. Δικαίω τίθεται το ζήτημα αυτό αλλά ζητάμε ουσιαστικά από τους Ευρωπαίους αγρότες να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και οι συνάδελφοι από τη Νέα Ζηλανδία ασχολούνται με τα ζήματα αυτά με τελώς διαφορετικό τρόπο. Αναφερόμαστε στη χρήση των γεών, στην ανταλλαγή γεών, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητούμε συγγνώμη για το τι προσπαθούμε να κάνουμε για τον προπολογισμό. Και θα ήθελα να βασιστούμε σε αυτή την πρόσφατη έρευνα και να δούμε πραγματικά τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τη γεωργία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 Ποια είναι η άποψη των κρατών μελών για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίως ε, το κομμάτι της γεωργίας, του πλαισίου αυτού. Εμείς ε, επιθυμούμε ή ευχαριστούμε καταρχήν για την υποστήριξη που μας προσφέρετε ως Επιτροπή, που προσπαθείτε να επιταχύνετε όσο δυνατόν περισσότερο τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ίδιο επιθυμεί διακαώς και η Κομισιόν. Και γι' αυτό το λόγο πριν από λίγες ημέρες ε, καταθέσαμε επικαιροποιημένους αριθμούς Νομίζω τους έχετε πάρει εντωμεταξύ. Είμαστε ευγνώμονες ε, που μας στηρίζετε ε, στην προσπάθειά μας επιτάχυνσης της ε, διαδικασίας. Αυτά που ακούσαμε από την Κυπριακή Προεδρία μας καθιστούν αισιόδοξου, διότι οι Κύπροι επιθυμούν διακαώς να προχωρήσουν τα πράγματα και το φθινόπωρο να έχει λάβει συγκεκριμένη μορφή η όλη συζήτηση. Ε, μονομένα μέλη αυτής της Επιτροπής ε, διερωτήθηκαν κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ε, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει η στιγμή να μιλάμε για ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν λάθος μήνυμα, γιατί πολλοί θα πίστευαν ότι εγκαταλείψαμε την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Και κατά τα άλλα, υπάρχει η δυνατότητα μέχρι το τέλος του σε να ολοκληρωθεί το θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και η γεωργική μεταρρύθμιση ακριβώς όπως προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2014. Άκουσα πάρα πολλές απόψεις ε, για την ερμηνεία της πρότασης του πολιτούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα ε, μεμονωμένα σχόλια για τις προτάσεις της Γεωργικής Επιτροπής, αλλά δεν ενδείκνυται σήμερα για μένα να τοποθετηθώ σε όλα αυτά. Το μόνο για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της επίτευξης συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν και με τον τρόπο αυτό να λάβει πλήρως υπόψη της τα συμφέροντα της Γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς την Επιτροπή, όπως και όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφής η θέση, έχει συζητηθεί και επανεπιβεβαιωθεί πολλές φορές αυτή την Επιτροπή. Στην Ολομέλεια ψηφίσαμε με ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτή λοιπόν ε, η σαφή θέση προέκυψε και από τους στόχους της Επιτροπής Σούρε, της έκθεσης Καρίγκα. Εμείς ε, επανειλημμένα έχουμε επιβεβαιώσει τη θέση μας στις διάφορες εκθέσεις, τις τελευταίες George Lyon και Albert Dess. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απολύτως αμφιβολία ότι παραμένουμε άκαμπτοι σε αυτή την κόκκινη γραμμή, στους όρους που θα πρέπει να διαπούν την ε, γεωργία. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις νέες ε, προκλήσεις. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε αγαπητοί συνέδελφοι, αλλά Νομίζω ότι πρέπει παρόλα αυτά να υπογραμμίσουμε και τις νέες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα οι γεωργοί γιατί βρίσκονται σε ένα τελείως διαφορετικό ανταγωνιστικό πλαίσιο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο απορρέει από την αστάθεια των διεθνών αγορών, είναι απότοκο ε, της ε, διακύμανση των τιμών, ε, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί ε, λόγω του ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές ε, μεταρρυθμίσεις από το Max Sharing μέχρι την, το θεματολόγιο του 2000 πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο και επειδή με τις συνθήκες της Λισαβόνας έχουμε αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες καλούμεθα να δώσουμε τη σωστή απάντηση σε μια γεωργία που όπως σας είπα βρίσκεται σε ένα νέο πλαίσιο. Κατόπιν τούτου, εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις ε, προτάσεις και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που εργάστηκαν με μεγάλη προσοχή και θέλω να Ελπίζω ότι θα λάβουν υπόψη τους ε, τις τροπολογίες. Ελπίζω και οι τροπολογίες κάπως να περιστούν σε ανθρώπινες διαστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπογραμμίσουμε ότι ο Γιωργός πρέπει ε, να βρίσκεται, να μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να ανταπεξέλθει και στις νέες δυσκολίε. Θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω ότι αυτά που μας είπε ο κύριος Λάιν στην αρχή βεβαίως ε, μπορούν να τροποποιηθούν από τις δικές σας ε, τι τροπολογίες που θα έχετε καταθέσει μέχρι το αργότερο 4 Σεπτεμβρίου 12 η ώρα. Θα πρέπει να έχουν φτάσει στη γραμματεία. Σας ευχαριστώ όλους και στο σημείο αυτό θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το σημείο υπαριθμών 5, το οποίο έχει άμεση σχέση βέβαια και με το προηγούμενο. Πρόκειται για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 13. Ε, και εδώ ε, η Έστερ είναι η συγγήτρια, Έστερ Ντελάγκε. Ε, έχει ε, γίνει αποδεκτή η έκθεση της Έσεντε Λάγκε σχετικά με την εντολή για την τριμερή συνάντηση και τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας του προπολογισμού. Το ε, Συμβούλιο θέλει να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή ημερομηνία. Εμείς καλούμεθα να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στην Έστερ για να παρουσιάσει την γνωμοδότησή της ε, και ε, θέλουν κατόπιν ενδεχομένω συνάδελφοι να παρέμβουν. Η Έστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο, ε, πριν τις θερινές διακοπές εντείνονται οι προσπάθειες και είπαμε ότι Ελπίζουμε η Κορεπέρ να είναι σαφής ως προς τις κατευθύνσεις ε, του Συμβουλίου και τελικά θα έχουμε στα τέλη Ιουλίου το αρμόδιο Συμβούλιο, λίγο αργότερα από συνήθως. Πάντως, ε, ακριβώς ε, η τελευταία χρονιά ενός πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου είναι και η πιο ευαίσθητη και μας το επισήμανε αυτό ο κύριος Λαβία. Έχουμε την πρόταση για αύξηση κατά 7% είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια δεν ε, διαφέρει αυτό τόσο τη γεωργία, γιατί εκεί προβλέπεται μόνο 2% αύξηση, ούτε καν φτάνουμε στο 2% για τη γεωργία, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, υπερήμερες πληρωμές που δεν είναι ακόμη γνωστές Επίσης, ε, από πολλές χώρες ασκούνται επικρίσεις για αυτή την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του προϋπολογισμού κατά 7%. Βέβαια το 0%, μηδενική αύξηση δηλαδή, ε, αντιλαμβάνεται και το Συμβούλιο ότι δεν είναι εφικτή. Ε, είχαμε αναλάβει πολλές υποχρεώσεις πληρωμών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τις στηρίσουμε και οι περισσότερες πληρωμές γίνονται προς το τέλος της περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών. Γι' αυτό δημιουργείται και πρόβλημα τώρα. Είχαμε ένα προπολογισμό με χαμηλό επίπεδο πληρωμών στην αρχή, οπότε ισορρέθηκαν οι πληρωμές για το τέλος, δεδομένης μεγάλης ανάληψης υποχρεώσεων που είχαμε φαίνεται ότι το Συμβούλιο ναι μεν προβλέπει νέες προτεραιότητες, αλλά δεν προβλέπει αντίστοιχη χρηματοδότησή τους με νέα κονδύλια. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία που μπορούμε να κάνουμε οικονομίες και σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Υπευλήθησαν αρκετές προτάσεις από τους συναδέλφους και επίσης από τους σκιώδεις συγητές για πιθανές οικονομίες από μερικά τμήματα του προϋπολογισμού. Και μάλιστα είναι γνωστά και κάποια στοιχεία της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων. Δεν θα επιβληθεί μια οριζόντια μείωση όπως σκεφτόμασταν πέρυσι, αλλά θα γίνει περιπτωσιολογική ανάλυση των δημοσιονομικών γραμμών. 8 εκατομμύρια φαίνεται θα φύγουν από τις διαφημίσεις, από τα μέτρα προώθησης, πολύ αφιβάλλω, γιατί θυμάστε πέρυσι είχαμε την κρίση με το ασχερίχια κόλλη, το εντεροβακτηρίδιο και ο Γερμανός Υπουργός ε, ε, καλύτερα να μην είχε μιλήσει γιατί με τις δηλώσεις του προκάλεσε τεράστια κρίση στον, στα απορροκυπευτικά ιδιαίτερα στα αγκουράκια και στις επέργειες. Οπότε δεν νομίζω να υπάρξει η μείωση του κονδυλίου της ε, προώθησης των προϊόντων, παρόλο που αυτό πρότεινε το Συμβούλιο κατά 8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ε, στηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θα πρέπει... Ε, να έχουμε από τη μια χιλιάδες παραγούς και από την άλλη ελάχιστες αλυσίδες διανομής που να ελέγχουν τις τιμές. Υπάρχει πρόβλεψη 35 εκατομμύρια για αυτό το θέμα το Συμβούλιο και 100 εκατομμύρια για την ανάπτυξη πέθρου. 300 εκατομμύρια θα πρέπει να βρούμε από την εκαθάριση των λογαριασμών. Πώς θα ανακτήσουμε όμως κονδύλια από το, το μέτρο αυτό. Είναι αρκετά φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. με τα 300 εκατομμύρια, όλα δε μάλλον το Συμβούλιο που συμφωνεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστική μια τέτοια πρόταση. Πού θα βρεθούν αυτά, από πού θα ανακτήσουν αυτά τα 300 εκατομμύρια. Και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, θα χρειαστεί και αύξηση των κονδυλίων. Πειραματικά σχέδια και προπαρασκευαστικές πράξεις. Η Επιτροπή Γεωργίας εδώ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κατά τη γνώμη μας ε, δεν έγιναν ε, σεβαστές ε, οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα ενημερωτική με πολλούς επισκέπτες, αλλά μιλούμε για τιμές και για αύξηση των τιμών σε επίπεδο καλλιεργιών, αλλά δεν μιλούμε για τα περιθώρια και για την κατανομή των περιθωρίων στις διάφορες αλυσίδες. Ένα Ολλανδικό Ινστιτούτο μας είπε ότι για ορισμένους τομείς, για τη χειροτροφία για παράδειγμα, διαπιστώνουμε 20-30% επενδύσεις, αλλά το στοιχείο που παίρνουμε από τις εκμεταλλεύσεις είναι αρνητικό. Και επίσης 10 με 15% έχουμε για τους παραγούς και 25 με 30% για τα σούπερ μάρκετ. Εκεί θέλουμε μία αλλαγή, μία επανισορρόπηση και είναι ανεπαρκή τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα άλλο πιλωτικό πρόγραμμα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο κύριος Μίλντερ είχε υποβάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έτυχε θερμής υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ε, έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια έρευνα για το, τα αντικειμενικά κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να μπουν οι πληρωμέ ένα εκτάριο στο ενιαίο το ομοιόμορφο μοντέλο. Αλλά δυστυχώ δεν έγινε αυτή η μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσαμε για περιφερειακές ενισχύσεις. Μας είπαν ότι οι ίσες πληρωμές δεν είναι κατά ανάγκη και δίκες, αλλά ζητήθηκε έρευνα για τα αντικειμενικά κριτήρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που δεν έγινε. Έχουμε μία πρόταση επίσης που υποστήριξαν όλες οι ομάδες, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι αγορές γίνονται όλο και πιο μεταβλητές και μάλιστα υπάρχουν στους πανεπιστημιακούς κύκλους γνώσεις για το πώς αποφύγουμε αυτές τις μεταβολές. Οι μεγάλοι σοκολατοπαραγωγοί, για παράδειγμα, ε, αγοράζουν ζάχαρη 1,5-2 χρόνια πριν αλλά η παραγωγή πώς θα, προετοιμαστούν για τα νέα μέτρα και τους νέους μηχανισμούς. Και μάλιστα, ενώ δεν προβλέπουμε αύξηση του γεωργικού προϋπολογισμού, ζητούμε τεράστιες προσαρμογές και θυσίες από τους γεωργούς. Επίσης, έχουμε τα άρθρα 21 και 24 του κανονισμού. Για τις ενημερωτικές εκστρατείες. θα πρέπει να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη αν όντω εφαρμόζουν ε, αυτά τα άρθρα 21 και 24, αν τα χρησιμοποιούν για την κατάρτιση, ε, ε, για, την ενημέρωση και τις γνωμοδοτήσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ ενθουσιασμός για τα θέματα αυτά. Οπότε χρησιμοποιούνται αυτά τα άρθρα από τα κράτη-μέλη για να ενημερωθούν οι παραγωγοί για τη μεταβλητότητα των αγορών. Όχι. Μόνο ένα κράτο μέλο χρησιμοποιεί αυτά τα άρθρα και μάλιστα με ανεπίσημο, με άτυπο τρόπο, παρόλο που το θέσαμε ω προτεραιότητα τη Επιτροπή Γεωργίας. Να ενημερώνουμε δηλαδή τους γεωργού ότι θα ε, λάβουν λιγότερα κονδύλια και να ενημερώνονται για τη ρευστότητα αυτή που επικρατεί στι αγορές. Ίσως ε, μία χώρα μόνο έβλαβε κάποια μέτρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, η, κατάθεση, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, λίγο πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, 23 Ιουλίου λίγη προθεσμία. Περιμένω τις προτάσεις σας, αλλά αναμένεται ένα σχετικά λιτό και φιδωλό δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε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 έχει καθυστερήσει λιγάκι όσον αφορά τη διαδικασία του προεπλογισμού. Έτσι λοιπόν, η τριμερή συνάντηση που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί για τον προεπλογισμό είχε από τη μία πλευρά ε, το κοινοβούλιο το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και από την άλλη πλευρά ήταν το Συμβούλιο το οποίο εκφράστηκε ε, σε καθαρά τεχνικό επίπεδο όμως ε, δεν είχε ούτε την ε, συγκεκριμένη άποψη της ε, Κοροπέρ ούτε του Συμβουλίου που προβλέπεται να εκδοθεί στο τέλος του μήνα. Αλλά πραγματικά μου φαίνεται λιγάκι περίεργο το ότι εμείς θα ολοκληρώσουμε τη φάση κατάθεσης τροπολογιών πριν να γνωρίζουμε ποια θα είναι η στάση του Συμβουλίου. Ίσως λοιπόν όλα αυτά να γίνουν πριν από τις 23, ε, να μας πει δηλαδή το Συμβούλιο ποια θα είναι η απόψή του. Νομίζω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως σας είπα, να κάνουμε εμείς δικές μας παρατηρήσεις, αφού θα έχουμε ακούσει την άποψη του Συμβουλίου. Και εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι η ανάγνωση που έγινε στις επιτροπές Προεπολογισμών σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, αυτή είναι μια πολύ περιοριστική ανάγνωση ε, και κατέληξε ε, σε ε, συμπέρασμα συμβιβασμός, εσωτερικός συμβασμός κάτι το οποίο όμως είναι πολύ αδύναμο ως θέση γιατί υπάρχει αντίθεση από τα, ανάμεσα στα κράτη που είναι καθαροί συνεισφορείς και στα άλλα που είναι καθαροί αποδέκτες. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η τεχνική ανάγνωση προσπάθησε να μετακυλήσει τις περικοπές σε άλλες τομείς, παραδείγματο χάρη ε, η πολιτική γειτονία. Ε, τα κονδύλια εκεί πραγματικά ε, περικόπηκαν τραγικά. Όπως και η 1α, έρευνα και καινοτομία για τους νέους, για την εκπαίδευση, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ από την άλλη, στην στον τομέα 2 που μας ενδιαφέρει εδώ πάρα πολύ, οι περικοπές είναι αρκετά επιλεκτικές. πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον με βάση αυτά που γνωρίζουμε να μας πει η Επιτροπή κατά πόσον οι προβλέψεις που γίνονται στο Συμβουλίο σχετικά με τις δαπάνες για την παρέμβαση στην αγορά, κατά πόσον τα κονδύλια αυτά θα είναι ικανοποιητικά ή κατά πόσον οι προβλέψεις του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα περιοριστικές. Και κάτι άλλο θέλω να πω, που έχει σχέση με, γενικότερα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο, διότι σήμερα το πρωί είδα ένα συμβούλιο το οποίο δεν έδειχνε να είναι ούτε καν διαθέσιμο να συζητήσουμε το θέμα των, ε, της εκταμίευσης των κονδυλίων. Αλλά ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές και σε σχέση με το Γεωργία, ότι παλαιότερα είχαμε τα μεμονωμένα κράτη-μέλη τα οποία έκαναν τις προβλέψεις δαπανών και τις ε, ανάγκες τους, ανάγκες κονδυλίων. Κατόπιν είχαμε την Επιτροπή η οποία έκανε τις ε, περικοπές και κατόπιν ερχόντουσαν τα κράτη-μέλη τα οποία όμως δεν ήθελαν να εκταμιεύσουν τα κονδύλια τα οποία είχαν περικοπεί από την Επιτροπή. Μα αυτά είχαν ε, κάνει τι προτάσει, περικόπηκαν και μετά δεν ήθελαν να εκταμιεύσουν τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδοξο που είναι δύσκολο να σταθεί. Κατά τα άλλα, το επίπεδο δαπανών ε, στην ε, Επιτροπή την, στην πολιτική των κρατών μελών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και εγώ δεν θα ήθελα οι δαπάνες για τη γεωργική ανάπτυξη, τα κονδύλια αυτά, να περικοπούν και να αναχαιτιστούν από τις πληρωμές. Γιατί αυτό θα ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη Γεωργία και γενικότερα, ε, γενικότερα για την γεωργική πολιτική, στο σύνολό της. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο λοιπόν έχει ζητήσει η Έστερ για κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο το ζήτημα αυτών των ημερομηνιών. Κανείς όμως δεν θα θέλει να βρίσκεται εδώ πέρα φαντάζομαι στι 30 Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου μόνο ότι είστε όλοι πάρα πολύ συμπαθεί και εργατικοί προκειμένου να γράφουμε τροπολογίες και να προσπαθούμε να βρούμε συμβαστικέ τροπολογίες. Στο παρελθόν αυτό που είχαμε κάνει είναι ότι είχαμε υποβάλει τροπολογίε βάσει τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια προσαρμόσαμε τι τροπολογίε αυτέ σε περίπτωση των διαφορετικά τα νούμερα από το Συμβούλιο. Τώρα βασιζόμαστε στου αριθμού του Κορεπέρ που λογικά θα πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στην τελική πρόταση του Συμβουλίου. Συνεπώς μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες και η Γραμματεία θα τις προσαρμόσει στη συνέχεια εφόσον τα αριθμητικά δεδομένα του Συμβουλίου διαφέρουν από τα δεδομένα τα αριθμητικά του Κορεπέρ. Πρέπει να εργαστούμε έτσι γιατί οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή Προπολογισμών όπως ο κ. Λαβία θέλουν να ψηφίσουν εγκαίρως και προκειμένου, εσείς φταίτε, ναι, και προκειμένου να καταφέρουν να ψηφίσουν εγκαίρως στην Επιτροπή Προπολογισμών και να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσει, εμείς ως Επιτροπή που βάλει γνωμοδότηση πρέπει να ψηφίσουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε μία τέτοια ημερομηνία η οποία βέβαια βρίσκεται πριν την ημερομηνία έγκριση της θέση του Συμβουλίου. Το έχουμε κάνει και αυτό στο παρελθόν και η Γραμματεία γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τις υποθέσεις. Ευχαριστώ. Bene, adesso Ulrich. Ευχαριστώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη συνάδελφο Έστερ Ντελάγκε διότι η συνάδελφος και το ταμπεραμένο της είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να αντιπαραβάλουμε στο Συμβούλιο. Γιατί πραγματικά με τρομάζει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το Συμβούλιο. Και διαπιστώνω ότι ε, στα εύκολα παρώνει το Συμβούλιο, αλλά όταν φτάνουν τα δύσκολα εξαφανίζεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι απαράδεκτο το ότι οι ε, πρόοδοι των πωλήσεων και ενώσει ε, παραγωγών θα πρέπει να υποστούν περικοπές. Ειδικά στις οργανώσεις των παραγωγών έχουμε συζητήσει επανειλημμένα ε, εδώ στην Επιτροπή μας το πώς είναι δυνατόν οι ενώσεις ε, παραγωγών να μπορούν να είναι ενωμένες και να αντιμετωπίσουν το λιανικό εμπόριο. Εδώ λοιπόν το να προβούμε σε περικοπές, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να ενδώσουμε σε αυτές τις ε, προτάσεις περικοπών. Ε, τα πιλωτικά προγράμματα, ε, τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ε, εξυπηρετούν τους γεωργούς και οι γεωργοί κάποια στιγμή θα μπορέσουν να παραιτηθούν από οποιασδήποτε μορφής, μορφή επιδότησης. Κατά τα άλλα, συνοπτικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτά τα κοντήλια στον προϋπολογισμό ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση του και σχετικά με τη μεταρρύθμιση όλοι εμείς ε, που πληττόμεθα από τις αλλαγές, η ε, Γεωργοί και όλοι οι άλλοι, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οφείλουμε να έχουμε έναν υγιή προπολογισμό. Ε, είμαστε σε καλά χέρια στην κυρία Ντελάνκε και αν μπορώ να τη στηρίξω ε, θα συνεχίσω να το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε και να δούμε τελικά πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε. Ευχαριστούμε Ουρίκ, George Λάιν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και ο συνάδελφος Τζοβάνι ε, Λαβία, και εγώ πολλές φορές ε, μπερδεύομαι και εντυπωσιάζομαι από τον τρόπο που χειρίζεται τα ζητήματα αυτά το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ο κύριος Λαμασούρ μας είχε πει ότι α, ε, όντως πρόκειται για ένα παιχνίδι μεταξύ ανθρώπων που ψεύδονται και νομίζω ότι α, ε, ήταν πολύ σαφή στο χαρακτηρισμό του αυτό. Έχουμε λοιπόν έναν προπολογισμό αυτή τη στιγμή που βασίζεται σε διαχειριστικέ αρχέ των κρατών μελών και των εκτιμήσεων που έχουν κάνει όσον αφορά τι μελλοντικέ δαπάνε που προβλέπονται στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου. Το Συμβούλιο λαμβάνει λοιπόν τι εκτιμήσει αυτέ, κόβει 20% γιατί θεωρεί ότι είναι υπερβολικέ και υπεραισιόδοξε και στη συνέχεια καταλήγει σε, ένα, σε μια πρόταση προπολογισμού. Ναι, 30% πολλέ φορέ είναι περικοπέ. Ο κύριο Λαβία μου λέει ότι οι περικοπές γίνονται πολλέ φορέ στην τάξη του 30%. Στη συνέχεια καταρτίζουν λοιπόν ένα προπολογισμό, ένα προβλεπόμενο προπολογισμό για το 2013 και έρχεται το Συμβούλιο τότε και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει φουσκώσει πάρα πολύ τα νούμερα. Αλλά ουσιαστικά στα δικά του τα νούμερα έχουν βασιστεί οι προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανάλυση αυτή που έγινε για συζήτηση μεταξύ ανθρώπων που ψεύδονται είναι πολύ καλή. Αυτό που θα ήθελα να μου πει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξή. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατά των ε, δαπανών και των περικοπών στι δαπανέ. Αρκεί αυτέ οι περικοπέ να μην έχουν πολύ αρνητικέ επιπτώσει όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Αν λοιπόν το Συμβούλιο προτείνει μειώσεις και περικοπές, δεν έχουμε δει βέβαια τις λεπτομέρειες, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των προτάσεων αυτού του Συμβουλίου. Ας μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και ποια είναι η άποψή τους όσον αφορά τις ε, περικοπές αυτές για την ε, χρηματοοικονομική υποστήριξη προς τον γεωργικό τομέα. Ποιε είναι οι προσδοκίε Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πού έγκυται τελικά που έγκυνται οι διαφορέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό α ακούσουμε την άποψη τη ε, Επιτροπή. Αλντολόγκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε κάπου, γιατί εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία θέση που μας δημιουργεί δυσκολίες και θα σε εξηγήσω γιατί. Εσείς ε, αναφέρεστε σε ένα προεπλογισμό ο οποίος κατά την άποψή μας είναι σωστός. Εντάξει, περιοριστικός, αλλά βασίζεται στη δική μας την ανάλυση των αναγκών, λαμβάνοντας ε, υπόψη, όπως είπε και ο κύριος Λαβία, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, προβλέψεις ή αν θέλετε τις ε, πληροφορίες που είχαμε πάρει από τα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι όσον αφορά τις ε, προβλέψεις των κρατών μελών, εμείς δεν είμαστε απόλυτοι, αλλά βασιζόμαστε σε μία μέθοδο στάθμισης. Σταθμίζουμε λοιπόν τις ανάγκες των κρατών μελών. Κυρίως όσον αφορά τη σύνταξη του προπολογισμού του 2013 είναι προφανές ε, ότι έχουμε λάβει υπόψη μας το phasing in των ε, ε, άμεσων πληρωμών η κοινή κυρική πολιτική λειτουργήσε αρκετά ικανοποιητικά γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε κάποιες παραδοχές δαπανών και επίσης θέλω να πω ότι σε αυτή την πρόταση προϋπολογισμού είναι σαφές ε, ότι ε, αναγκαστήκαμε να λάβουμε υπόψη μας κάποιες ε, θέσεις που είχαν με το health check το περίφημο. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη επιτάχυνση. Νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως. Πραγματικά επιταχύνθηκαν τα προγράμματα και από ό,τι φαίνεται, κατά τη διάρκεια του 2013 θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση. Άρα δηλαδή καθίσταται απαραίτητο ε, να παραμείνουν τουλάχιστον οι πιστώσεις πληρωμών. Λάβαμε υπόψη μας ε, την άποψη του Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι μας ανησυχεί και επίσης ε, αναλύσαμε και τις περικοπές τις οποίες προτείνει το Συμβούλιο, τις αναλύσαμε πολύ προσεκτικά για να προσπαθήσουμε να δούμε ε, τι μπορεί κανείς να κάνει με αυτές τις ε, περικοπές. Είναι σαφές ότι αυτά τα οποία προτείνονται σχετικά με την clearance είναι αυθαίρετα. Δεν βασίζονται πουθενά. Αυτά τα 300 περίπου 20 εκατομμύρια για μας είναι μια τελείως αυθαίρετη, ένα τελείως αυθαίρετο ποσό. Επίσης, μας ανησυχούν και άλλα θέματα που προφανώς ε, αυτή τη στιγμή εμείς ε, θεωρούμε ότι ε, τα θέματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις προβλέψεις μας. Έτσι λοιπόν οι παράμετροι που είχαμε προτείνει εμείς στην πρόταση προπολογισμού παραμένουν οι ίδιες και προφανές είναι ότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να αναθεωρήσουμε κάποιες θέσεις μας. Είναι σωστό αυτό που είπε ο συνάδελφος κύριος Λαβία και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Ντελάγκε. Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον, νομίζω το Σεπτέμβρη, θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην διορθωτική επιστολή που θα σας σταλεί ε, τον Σεπτέμβριο. Να αρχίσουμε να δουλεύουμε τον Οκτώβριο. Εκεί θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τις αρχικές παραδοχές με βάση δηλαδή αυτές που, που καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό. Και ίσως τότε πια θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με την πρόταση που έχει κατατεθεί σήμερα στο Συμβούλιο. Εγώ προφανώς ε, πρόεδρε είμαι ανοιχτό σε, σε απόψεις ε, και θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προφανώς της εισηγήτριας, ε, της κυρίας Ντελάνγκε, να έχουμε, γιατί όχι, μια πιο ουσιαστική συζήτηση για τις ε, προτάσεις του Συμβουλίου. Και αν θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε και τη δουλειά ε, χωρίς καθυστερήσεις ε, για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Θα ήθελα τώρα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ λιγάκι στα πιλωτικά προγράμματα. Εδώ πρόκειται για ένα στοιχείο που έρχεται και επανέρχεται ε, στις συζητήσεις μας, τουλάχιστον αυτή την εποχή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο στα πιλωτικά προγράμματα και σε προκατακτικές δράσεις ως ένα εργαλείο πολιτικής πράξης. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλές μελέτες που σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, υπάρχει περίπτωση να καπελώσουν τα πιλωτικά προγράμματα και γι' αυτό το λόγο ανησυχούμε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρχουν επικαλύψεις ε, ανάμεσα στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτών που έχουμε ήδη πράξει ή που πράττουμε αυτή τη στιγμή. Σε γενικέ γραμμές, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι μια πιο τεχνική συνάντηση, συζήτηση θα μπορούσε, θα μας επέτρεπε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα των πιλωτικών προγραμμάτων που έχουν προταθεί από τα κρατημέλη τόσο κατά το παρελθόν όσο και τώρα. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ντελάγκε να μας δώσει τη δυνατότητα να μπούμε περισσότερες σε λεπτομέρειες αυτών των προγραμμάτων. Θα ήθελα όμως να τοποθετηθώ και σε ορισμένα θέματα ε, τα οποία ε, λέχθησαν σήμερα το πρωί από την κυρία Ντελάγκε απλά και μόνο για να διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία ε, τα οποία έχουν πάντα σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα. Όπως σας είπα λοιπόν, κατά το παρελθόν όσον αφορά στη μελέτη περιθωρίου και τιμών Είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες που κατά την άποψή μου ανταποκρίνονται σε αυτά που μας ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το πιλωτικό πρόγραμμα. Ένα, υπάρχει ένα εργαλείο παρακολούθησης ε, περιθωρίων και τιμών και εμείς σκεφτήκαμε ότι αυτό που είναι πραγματικά απαραίτητο κύριε Πρόεδρε και κυρία Ντελάνγκε, είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων και να ε, δώσουμε τη δυνατότητα ε, στην κοινή γνώμη να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά ε, να γίνουν κατανοητά ως μια ε, χειρονομία καλής θέλησης για να ανταποκριθούμε σε αυτά που μας ζητάτε. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις που αφορούν στα περιθώρια γιατί νομίζω ότι ελέγχθη αυτό σήμερα, υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Εμείς έχουμε πολύ καλές μελέτες που αφορούν στα αγροτικά περιθώρια και δεν έχουμε τόσο ασχοληθεί με τα περιθώρια του κάθε τομέα. Θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε με την κυρία Ντελάνγκε για να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ή δυνατόν από κοινού να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Πρόεδρε, Μπορούμε βέβαια να μπούμε και σε λεπτομέρειες και στα άλλα πιλωτικά προγράμματα, αλλά σας είπα, θα προτιμούσα όλα αυτά να γίνουν στο πλαίσιο μια τεχνική συνάντηση σε διμερές επίπεδο ε, και όσον αφορά και το σχέδιο του κυρίου Μούλντερ. Ε, ε, το Είμαστε τώρα λίγο πριν από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχουμε 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη που έχει προβλεφθεί. Όσον αφορά τώρα την διακύμανση των τιμών, να μπορούν οι γεωργοί να γνωρίζουν καλύτερα αυτή την διακύμανση. Πράγματι κύριε Πρόεδρε, αυτό το στοιχείο ε, μαζί με την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να εξεταστεί για να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Και ξέρετε γιατί. Γιατί κάθε τομέας έχει την δική του την προϊστορία. Υπάρχουν οι αγορές οι οποίοι σε σχέση με τη διακύμανση των τιμών ε, συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά. Αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω με τον κατάλογό μου, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο και γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Αλντολόγκο και τώρα... Για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Έστερ και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η Έστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα προφανώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση που μας έδωσε. Νομίζω ότι συμφωνούμε για πολλά, σε πολλά σημεία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί μαζί μας όσον αφορά το ζήτημα της καθάρισης των λογαριασμών. Και βλέπουμε ότι το Συμβούλιο όντω έχει λειτουργήσει πολύ επιλεκτικά σε κάποια σημεία, έχει μια πολύ επιλεκτική προσέγγιση. Νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο οι σκιώδεις ε, εισηγητές να συμμετέχουν και αυτοί σε κάποια συζήτηση που θα πρέπει να κάνω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε αν θα γίνουν κάποιες ε, αλλαγές. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία όντως θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε ή να τροποποιήσουμε. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, νομίζω ότι επιμακρών θα πρέπει να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Και ο κύριος Μούλντερ μου είχε πει το 2009 ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε προτείνει να εξετάσουμε τα κριτήρια της ε, κατανομής ε, του επιδόματος εισοδήματος, της ενίσχυσης εισοδήματος. Και νομίζω ότι όταν τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία το 2011 ήταν πια πάρα πολύ αργά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Βλέπουμε ότι έχει υπογραφεί μια σύμβαση και ουσιαστικά χάνουμε πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ προ αυτό, προ τα αντικειμενικά κριτήρια. Τώρα, όσον αφορά τα περιθώρια, και αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πάντω πάρα πολύ με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που από ό,τι φαίνεται επιθυμεί να συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να επέλθουν κάποιε βελτιώσει. Η κυρία Μαγκίνε αναφέρθηκε σε μια άτυπη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Μάλιστα είναι επικεφαλής μιας άτυπης ομάδας διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε περισσότερο για τα περιθώρια, τις τιμές, σε ένα ευρύτερο όμως επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δούμε αν μπορεί να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία το σύστημα το οποίο έχουμε. Εγώ ευχαρίστως θα συμμετείχα σε μια τέτοια συζήτηση. Όσον αφορά τώρα τη μεταβλητότητα, Καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπατε, ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης. Το ότι υπάρχουν όμως οι εναλλακτικέ αυτές δεν σημαίνει ότι θα τις χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ή ότι θα καταφέρουν να τις χρησιμοποιήσουν προς το συμφέρον των γεωργών και της γεωργικής πολιτικής. Και αυτό το επίπεδο μας μας ενδιαφέρει. Όταν λέτε ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές και να γίνει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, Θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό να απασχολήσει και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει σαφώς να αντλήσουμε όποια θετικά διδάγματα υπάρχουν από τις βέλτιστες πρακτικές. Ενδεχομένως, βέβαια, να είναι πολύ αργά προκειμένου να επέλθει κάποια βελτίωση αυτή τη στιγμή για τον προπολογισμό, αλλά μη τι άλλο θα πρέπει οι γεωργοί να ενημερωθούν για τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια του 21ου αιώνα. και ξέρετε ότι υπάρχει και μία οριζόντια ανώτατη τιμή για τις ε, επιδοτήσεις οι οποίες προβλέπονται. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κονδύλια από το EFSF, EF, EFS, e με συγχωρείτε, για κάποια προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα διαβίου μάθησης και κατάρτισης. Και ενδεχομένω θα μπορούσε να γίνει μια κάποια μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές Ενδεχομένως από το κοινωνικό ταμείο θα μπορούσαν να προέλθουν τα χρήματα αυτά. Πάντως ελπίζω να μπορούμε να συναντηθούμε ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Πολύ ωραία λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ας μην ξεχνάμε για άλλη μια φορά καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών 23 Ιουλίου 12 η ώρα. Τώρα λοιπόν πάμε στο σημείο υπαριθμών 6 της ημερήσιας ε, διάταξης ε, που νομίζω ότι μπορούμε να το εξετάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για την ε, μισό λεπτό για την πρότιση των γεωργικών προϊόντων. Ε, πρόκειται για την τροπή του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τι ενέργειε ερμηνεία και πρόθεση υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στι τρίτε χώρε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ζωζέ και νομίζω ότι ήρθε και ο διευθυντή Πατσάκοβιτ. Ο Ζωζέ έχει το λόγο. donc effectivement c'est un Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω πρόκειται για ένα σχέδιο εκθέση που αφορά θέμα ευθυγράμμισης. Είναι ε, σχετικά απλό, ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο έχει την ευθυγράμμιση του κανονισμού της 10 της Δεκεμβρίου ε, του κανονισμού 3-2008 σχετικά με ενέργειες ενημέρωση και προώθηση υπέρ των γεωρικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες και ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια κατανομή που σέβεται το πνεύμα της συνθήκης μεταξύ των γενικών διατάξεων και των ε, ειδικών. Έχουμε το άρθρο 290 καταρχήν, τα πιο γενικά και τα πιο τεχνικά θέματα στο άρθρο 291. Αυτά τα δύο άρθρα της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν εδώ. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες που ενισχύουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το κατάλογο των θεμάτων και προϊόντων που είναι επιλέξιμα για τις ε, δράσεις πρόθεσης, γιατί στόχος μας είναι πραγματικά να ενισχύσουμε και να δώσουμε μια πιο οριζόντια ε, άποψη και στη θέση και στη διατύπωση. Βλέπετε το κατάλογο θεμάτων και προϊόντων που επισυνάφθηκε στη βασική πράξη με τη μορφή παραρτήματος για να είναι πιο σαφή τα πράγματα. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, βλέπω ότι κάποιοι συναδελφοί έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν, αλλά νομίζω ότι ε, θέλουν περισσότερο να μιλήσουν για την επόμενη έκθεση. Έτσι δεν είναι. Ο Δόκτωρ Πασέκο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως θέλετε το λόγο, είπατε ότι ενδιαφέρεστε. Παρακαλώ κύριε Πασέκο. Ευχαριστώ, θα είμαι και εγώ λακωνικότατος. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μποβέ για την έκθεσή του γιατί νομίζω ότι για τα ουσιώδη είμαστε σύμφωνοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μα ενδιαφέρει πολύ η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανέβρεση Λύση. Σε ό,τι αφορά τι λεπτομέρειε, θα τι αφήσω για το επόμενο θέμα. Εμεί. Ε, προτιμούμε μεγαλύτερη ελαστικότητα σε κάποιες τροπολογίες, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Άλλο, ο Ζωζέ, θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, ωραία, τέλεια. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, στο 8 τη ημερήσιας διάταξης, λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές, μισό λεπτό, το 7 λέει ο πρόεδρος, ε, ε, έκανα λάθος, ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και πρόθεση τους, μια στρατηγική για την πρόθεση των γεύσεων της Ευρώπης. Ο Ζωζέ Μπούβε είναι εισηγητής και μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, στις 30 Μαρτίου ε, έχουμε την ε, γνωμοδότηση του κ. Μπούβε για τις γεύσεις στην Ευρώπη. Αυτό εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου του 2012, αλλά θέλουμε όμως να υπάρχει μια πιο ουσιαστική τοποθέτηση και γι' αυτό δίνουμε το λόγο σε εσένα, Ζωζέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Όντως, στόχος μας στην έκθεση αυτή είναι να βασιστούμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου του 2012 όσον αφορά την πρόθεση και την ημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα. Θεωρώ ότι την ανακοίνωση αυτή είναι πολύ θετική, κατευθύνεται σωστό δρόμο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να συμβάλλει στο ότι τα μέσα προώθησης ε, δεν βασίζονται μόνο στα βασικά γεωργικά προϊόντα, αλλά και στα τρόφιμα ποιότητος και σε αυτά τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο περιμένει ο καταναλωτής, ο Ευρωπαίος ε, πολίτης, το βλέπουμε αυτό και σε αναλύσεις του Ευρωβαρομέτρου, είναι να διαθέτουν τοπικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητος, προϊόντα τα οποία μπορεί, να μπορεί εύκολα να γνωρίσει ο καταναλωτής. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει η γενική προσέγγιση να είναι πολύ πιο σαφής, πολύ πιο επιλεκτική και ένα πρώτο στάδιο θα πρέπει να είναι ενδυνάμωση τη συνεκτικότητα των δράσεων και μια συνέργεια μεταξύ διαφορετικών μέσων πρόθεση που υφίστανται. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποια πολύ σαφή στοιχεία όσον αφορά την πρόθεση των ποιοτικών προϊόντων. Αυτά τα μέσα θα πρέπει να έχουν να κάνουν με την προέλευση, τη γεωρική προέλευση των προϊόντων, με τον τρόπο παραγωγής τους, με τον τρόπο καλλιέργειάς τους και ότι θα πρέπει να υπάρχει το κλασικό καθεστώς προστασίας τους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να προωθηθούν περισσότερο τα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγονται και προϊόντα τοπικά. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν, δεν είχε τονιστεί ποτέ στο παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδεικνύουν τελικά ότι οι τρόποι παραγωγής συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών αγορών και στην πρόθεση των τοπικών προϊόντων και ότι κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν περισσότερο στην βιοπικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντο. Και θα πρέπει να φαίνεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται προστιθέμενη αξία για του γεωργού σε τοπικό επίπεδο. Ανάμεσα στι προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία και το στοιχείο αυτό και τα μέσα αυτά θα πρέπει να υφίστανται προκειμένου να προωθηθεί η γεωγραφικά εντοπισμένη γεωργία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βέβαια αυτοί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ένας νέος πιο σημαντικός προπολογισμό στα σχετικά μέτρα προώθησης και ενημέρωσης. Πριν από λίγο μιλήσαμε για το ζήτημα του προπολογισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό, ξεκάθαρο προπολογισμό που θα εξυπηρετεί όλους τους στόχους μας, αλλά όχι με οποιονδήποτε τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Έχουμε διάφορους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Κυρία Πατράου Νέβες πρώτα και μετά η κυρία Γιούζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι τεράστια αυτή η ευκαιρία που έχουμε, μοναδική, για να αισθανθούν, να αισθανθούν επιτέλους οι γεωργοί ότι όλε οι προσπάθειε του και όλε οι υποχρεωτικέ επενδύσεις που έκαναν για τη δημόσια υγεία, για το περιβάλλον, για την ευημερία των ζώων και για τι ε, κοινωνικέ συνθήκε όσων ε, καλλιεργούν τη γη, ότι όλες αυτές οι προσπάθειες άξαν τον κόπο και έχουν ένα αντίκρισμα. Αν η συμμόρφωση με τις πιο απαιτητικές προϋποθέσεις ε, για τη γεωργία δεν δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία των προϊόντων και δεν αυξήσουν τα εισοδήματα των γεωργών, τότε θα μείνουμε μόνο με ένα, με ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Θέλουμε να προωθήσουμε τη γεωργική μας παραγωγή, αλλά θα έλεγα σε τοπικό επίπεδο, σε αγορές εγκύτητας, με ε, στενά κυκλώματα, αλλά και σε, σε επίπεδο νέας αγοράς να δώσουμε έμφαση στον ενιαίο χώρο χωρίς σύνορα με 500 εκατομμύρια καταναλωτές και φυσικά σε τρίτο επίπεδο στην παγκόσμια αγορά ε, όπου θα είμαστε ανταγωνιστικοί με ποιότητα ε, και ποικιλία. Η πρόθεση ποιοτικών προϊόντων δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσουμε ε, γερή θέση στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε κάποια προγράμματα πρόθεσης. Πάντως Πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει η πολιτική προαγωγής αυτών των προϊόντων να ε, στηρίξει τους Ευρωπαίους παραγωγούς, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν την αύξηση της κατανάλωσης σε αναδυόμενες οικονομίες. Γιατί ε, οι εξαγωγέ θα γίνουν όχι μόνο σε νέε αγορέ, με τι εξαγωγέ βελτιώνεται και η κατάσταση των επιχειρήσεων και δημιουργούνται και θέσει απασχόληση. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να δημιουργήσουν συνεταιρισμού, ομάδε, ώστε να δημιουργήσουν μια κρίσιμη μάζα μεταξύ του για να μπορέσουν να έχουν μια παρουσία στο διεθνέ εμπόριο, κάτι που μέχρι στιγμή ήταν δύσκολο. Να διευκολύνουμε τη διευθέτηση προβλημάτων που αφορούν τι αγωγέ και να παράσχουμε στους εισαγωγείς ε, ενημέρωση και ίσως να έχουμε και μια κεντρική θεματολογική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή την άποψη καλό θα ήταν να δίνουμε στοιχεία για τις εξαγωγές, να δίνουμε πληροφορίες για επαφές, χώρες, προς ανατολισμούς των εξαγωγών σε όλους και χονδρέμπορους και ε, λιανέμπορους Επίση, μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιε εκστρατείε ώστε να εθαρρύνουμε τι οργανώσει, ε, τι επαγγελματικέ οργανώσει των κρατών μελών να δραστηριοποιηθούν ώστε να υποβάλουν υποψηφιότητα σε προγράμματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, σε προγράμματα που συμμετέχουν πολλέ χώρε. Δυνατότητα να προωθήσουμε και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Επίσης με τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ε, εφαρμογή, με τη συμμόρφωση με τις ε, απαιτήσει ε, για την υγειονομική ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα, τις αυστηρές προϋποθέσεις για το περιβάλλον, την ευημερία των ζώων, τα, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ώστε αυτές οι απαιτήσει και οι προϋποθέσεις που επιβάλλουμε στους δικούς μας γεωργούς να αξιοποιούνται και να δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία και στην εξωτερική αγορά. Γιατί κάνουν που κάνουν τι θυσίε του. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν αντίκρισμα. Επίση, ε, χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη διαφάνεια στην επιλογή των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς για τα κράτη-μέλη. Αξιολόγηση των προγραμμάτων. Και αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Θα πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση με συγκεκριμένου δείκτες. Για παράδειγμα, η αύξηση του μερίδιου τη αγορά είναι ένας σαφή αντικειμενικό δείκτης. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι δείκτες που να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των προγραμμάτων. Επίση, ό,τι αφορά την παρούσα πολιτική ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων. Είχαμε μερικά αίσια αποτελέσματα μέχρι στιγμή στην πολιτική αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κάποια απλούστευση και κάποια βελτίωση ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άκθος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, ο εισηγητή μα ήδη το επισήμανε ότι είναι κρίσιμο αυτό το θέμα του προπολογισμού και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και την πιθανότητα υψηλότερων προκαταβολών για ορισμένε επαγγελματικέ οργανώσει. 50% αντί για 30% προκαταβολή όπως προτείνεται και τέλος θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα τον εισηγητή μας για την έκθεση πρωτοβουλίας ε, την οποία προσυπογράφω ως προς τις αδρές γραμμές της. Τώρα, λόγω της, του περιορισμού στις σελίδες που έχουμε δεν μπορέσαμε να είμαστε πιο διεξοδικοί σε ό,τι αφορά αυτή τη μια όχι μόνο μιας γεωργίας που θα εξασφαλίζει την επισητιστική ασφάλεια και την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, αλλά που θα είναι ταυτόχρονα ικανή να εξασφαλίσει ένα δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς. Αυτό το σημείο θα πρέπει οπωσδήποτε να το τονίσουμε και στην έκθεση αυτή. Είμαι φυσικά στη διάθεση του εισηγητού για συνεργασία για όλα τα σημεία που ανέφερα και πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε για να είναι πιο ικανοποιητική έκθεση, κυρίως σε αυτούς που έχουν υψηλές προσδοκίες ε, από εμά και που είναι οι γεωργοί μας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατραονέβες. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε καλύτερα να περιστούμε λιγάκι για να έχουμε και συνεδρίες των συντονιστών. Αγιούζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι επιγραμματική. Νομίζω ότι είναι μια ε, πραγματικά μοναδική ευκαιρία για μια ουσιαστική στρατηγική προώθηση των γεωρικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι σημαντικό και για την ε, φήμη των ε, κοινοτικών προϊόντων και εντός και εκτός της κοινοτικής αγοράς. Θα πρέπει να δοθεί έφταση στη βιοπικιλότητα, στην παράδοση, στις υψηλές προδιαγραφές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία, την προστασία περιβάλλοντος, ευημερία των ζώων και ούτω καθεξής. Πολλές φορές στην έκθεση γίνεται ε, συγκρίση και αναφέρονται τα στενά κυκλώματα ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Συμφωνώ και το περιέλαβε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Τέτοιου είδους προώθηση των αγορών εγκύτητας και των ε, μικρών κυκλωμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, βιώσιμη καλλιέργεια. Αλλά στην Ευρώπη όλες οι καλλιέργειες είναι βιώσιμες. Ε, εδώ έχουμε τι πιο βιώσιμε καλλιέργειε από όλο τον κόσμο. Οπότε ίσω δεν είναι και πολύ εύστοχη αυτή η αναφορά. Φαντάζομαι εννοείται την οικολογική καλλιέργεια ή την ολοκληρωμένη καλλιέργεια. Και αυτό όμω εμπίπτει στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Επίση, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθηθούν τα γεωργικά προϊόντα που δίνουν ε, στο πρόγραμμα μια πραγματικά προστιθέμενη αξία και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Και εδώ δίνουμε έφαση στα προγράμματα ονομασίας προέλευσης, γεωργικές ε, έδειξει κτλ. Αλλά όχι αποκλειστικά σε αυτά εμποδίζοντας την πρόθεση και άλλων προϊόντων. Επίσης, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε σημεία που πραγματικά βελτιώνουν την πολιτική πρόθεση στο γεωργικό προϊόντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να προωθούνται προτάσεις μεταξύ πολλών κρατών μελών που θα καλύπτουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Ε, να χρησιμοποιούμε και το σήμα, να απλουστεύεται η διαχείριση των προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων με πολλές χώρες και να δίνεται τεχνική υποστήριξη στις ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ό,τι αφορά τις στρατηγικές τους για το μάρκετινγκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Πόλσον και μετά κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τον κύριο Μποβέ. Ναι, μία μικρή περιφερειακή αλυσίδα διανομής, αυτό είναι όντως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όντως πολλές γεωγραφικές ζώνες στην Ευρώπη, όπου για καθαρά φυσικούς λόγους οι εκμεταλλεύσεις γεωργικές είναι πολύ μικρές και οι ζώνες αυτές βέβαια απέχουν πολύ από τις μεγάλες αγορές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες αλυσίδες διανομής προκειμένου όλοι να λειτουργούν σωστά. Η λεπτομέρεια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όταν όμως μιλάμε για τοπικές αγορές και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε τοπική παραγωγή, θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου πάντα ότι ήδη σήμερα άνω του 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε περιοχές οι οποίες είναι πυκνοκατοικημένες Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ετικετοθεσία προκειμένου να μας σε θέση να βλέπουμε ποια είναι η προέλευση των προϊόντων. Επίσης, υπάρχουν δύο ακόμα στοιχεία τα οποία ενδεχομένω να μην έχουν να κάνουν με τη διάθεση στην αγορά των γεωργικών προϊόντων, αλλά είναι εξίσου σημαντικά. Από τη μια, θα πρέπει να διατηρήσουμε τα παραδοσιακά προϊόντα, καθώς επίσης και την παραδοσιακή προπαρασκευή παραγωγή των προϊόντων. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες συγκεκριμένε γνώσεις που υφίστανται όσον αφορά την παραγωγή ποιοτικών διατροφικών προϊόντων. Ξέρετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η παραγωγή των τροφίμων γίνεται με τρόπο πολύ πιο βιομηχανοποιημένο και ψηφιακό σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε και την τοπική βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων. Αν χαθούν οι γνώσεις αυτές, τότε η μελλοντική γενιά δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτές τις γνώσεις ή να τις ψηφιοποιήσει, αν θέλετε. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι να φερθούμε στην ε, βιοπικιλότητα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, η βιοπικιλότητα δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα αυτό της ύπαρξης πολλών διαφορετικών άγριων ειδών. Όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα αναφερόμαστε ουσιαστικά και στην ε, υπεράσπιση κάποιων ε, τοπικών περιφερειακών ειδών, ζώων και φυτών. Η προϋπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε μία, ένα πολύ καλό επίπεδο γεωργίας για το μέλλον. Να καταφέρουμε δηλαδή να διασώσουμε την μελλοντική γεωργία. Θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα στο μέλλον. Η Γκαρσία και μετά κύριος Καπόλα Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνική, τηλεγραφική και σύντομη κύριε Σιγητά. Εσθενίζομαι πλήρως ε, τα σχόλια της κυρίας Αγιούσο. Αλλήμωνο. Άλλωστε ήταν ε, ιδιαίτερα εύστοχη σε πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο τίνα. Για όλα τα είδη της παραγωγής και για όλους τους θύλακε ε, πρόθεσης που καλύπτονται από την αγροτική ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να προβλέψουμε εδώ κονδύλια, γιατί το πρώτο πρόβλημα που έχουμε με την έκθεση αυτή είναι ότι δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση των ε, κονδυλίων για τα μέτρα πρόθεσης. Οπότε, αν ε, παγώσει τα κονδύλια αυτά για την πρόθεση, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην περιορίσουμε εμείς ε, το πεδίο εφαρμογής, ώστε τελικά να, να είναι αναποτελεσματικά αυτά τα μέτρα της πρόθεσης. Αν υπάρχουν μέτρα που καλύπτονται από την αγροτική ανάπτυξη, να τα αφήσουμε εκεί. Επίσης, η ιδέα μας για την πρόθεση των ευρωπαϊκών προϊόντων θα πρέπει να έχει πολύ πιο υψηλές βλέψεις, όπως μας τόνισε και η κυρία Γιούσο. Κάτι άλλο που είπαν οι συνάδελφοι. Όλα τα προϊόντα που θεωρούνται τρόφιμα θα πρέπει με ίσες συνθήκες και χωρίς διακριτική μεταχείριση να συμμετέχουν στα μέτρα πρόθεσης. Στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που τα προϊόντα αυτά θεωρούνται τρόφιμα. Οπότε θα πρέπει να τονίσουμε αν τα μέτρα προωθηση κάποιων προϊόντων που, όπως ο ίνος που αυτή τη στιγμή περιορίζονται στη διεθνή αγορά μπορούν να επεκταθούν και στην εσωτερική αγορά. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη επέκταση. Το είπα και την προηγούμενη φορά και μάλιστα θα καταθέσω και σχετική τροπολογία. Και τέλο, κύριε Μποβέ. Φαίνεται ότι στο έγγραφο δεν αναφερθήκατε ιδιαίτερα στο ρόλο που μπορεί να παίξει η προώθηση σε συνθήκες κρίσης της αγοράς. Αυτό ελάχιστα το αναφέρεται ακροθυγός. Πιστεύω όμως ότι όχι μόνο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη ποιότητα, αλλά αυτή είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία να εφοδιαστούμε με ένα μηχανισμό που θα προστατεύσει τους γεωργούς και την ε, κοινωτική παραγωγή και από τις ε, κρίσεις. Ευχαριστώ ο κύριος Λουίς Καπόλα Σάντος και μετά Μάρκ Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ επιγραμματικός. Θα ήθελα εκ μέρους της πολιτικής ομάδας μου και εκ μέρους της και ηγετριά μας της κυρίας Βιτόρια Νταντζίλα που δυστυχώς καθυστερεί και θα αργήσει ε, να έρθει στις Βρυξέλλες. Θα έρθει σήμερα το βράδυ. Ε, δεν μπορεί να λάβει μέρο στη συζήτηση. Εκ μέρου πάντω και εκ μέρου ομάδα ήθελα να πω ότι εστερνιζόμαστε τι ε, κατευθυντήριε γραμμέ του εισηγητού μα, γιατί την ε, προηγούμενη φορά δώσαμε έφαση στην ποσότητα αντί στην ποιότητα και χαιρόμαστε που αυτή τη φορά γίνεται μια μεταστροφή και δίνουμε έφαση στην ποιότητα και στην προσεθέμενη αξία των κοινοτικών, προϊόντων. Έχω μια προσωπική ερώτηση προς τον εισηγητή. Μιλάτε για το τέλος των ενισχύσεων προς την πρόθεση όταν ε, θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μετά από σκάνδαλα διατροφικά ή επισητιστικά. Είδατε την περίπτωση του εντεροβακτηριδίου στην ε, Γερμανία και την αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος πολλών κοινοτικών παραγών. Σε τέτοιες περιπτώσεις δικαιολογούνται μέτρα πρόθεση για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης μετά από τέτοια σκάνδαλα. Θα ήθελα να το ξανασκεφτεί παρακαλώ ο εισηγητής, το απευθύνω έκκληση. Ίσως θα έπρεπε πιο διεξοδικά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Λουίς. Ο Μάρκ Ταραμπέλα και τελευταίος, κύριε Βάρκ. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι όντω είναι πολύ καλή η έκθεση του κυρίου Μποβέ, ιδίω όσον αφορά το ζήτημα τη ποιότητα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την κατανάλωση των τοπικών προϊόντων και όχι να προωθήσουμε ποιοτικέ βιολογικέ ντομάτε που έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε λοιπόν την τοπική κατανάλωση. Όσον αφορά επίση την βιώσιμη καλλιέργεια, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε καλλιέργειες βιώσιμες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε μία σειρά από τα οποία έχουμε υποστηρίξει και σε άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για παράδειγμα και ότι ε, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, αν θέλετε, όλες αυτές οι, όλοι αυτοί οι στόχοι μας κάθε φορά που ε, αναφερόμαστε σε ζητήματα όπως για παράδειγμα η κατανάλωση φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων στο σχολείο. Καθώς επίσης πρέπει να προωθήσουμε και την διασύνδεση, η οποία θα πρέπει ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί ανάμεσα στους γεωργούς και τους ε, πολίτες. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται και στη δική μου την περιοχή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εμβαθυθούν οι σχέσεις αυτές και αυτό θα μπορέσει να επηρεάσει την κατανάλωση προϊόντων τόσο από τα παιδιά, αλλά και από τα παιδιά αυτά τα οποία θα ενηλικιωθούν κάποια μέρα και ουσιαστικά θα επηρεάσει και την ε, συμπεριφορά γενικότερα στο οικογενειακό πλαίσιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία κύριε Ταραμπέλα Χάιουαρτ και μετά Μαγκίνη. Ω ηγητή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζωζέ Μποβέ για το κείμενο αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ομοιόμορφη στρατηγική όσον αφορά την πρόθεση και την ενημέρωση για τα γεωρικά προϊόντα. Και όντω μια τέτοια πολιτική όχι μόνο θα πρέπει να καταρτιστεί, αλλά θα πρέπει επίση να επιβραβεύει και του ε, γεωργού αυτού οι οποίοι με βιώσιμη τρόπο μπορούν να ανταποκριθούν στι νέε προκλήσει. Συμφωνώ επίση με του στόχου οι οποίοι ε, παρατίθενται εδώ πέρα, να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία, καθώ επίση και μια καλύτερη στρατηγική για την πρόθεση των πρόοδων αυτών και χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών μέσων. Η απλούστευση είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να έχουμε μια πολιτική προώθηση την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο γεωργοί όσο και οι καταναλωτέ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί στον προπολογισμό, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφτούν τα παρέτα κονδύλια για τη στρατηγική πρόθεση. Θα πρέπει ο σχετικό προπολογισμό να αυξηθεί όπως άλλωστε λέει και ο εισηγητή, και θα πρέπει οι καταναλωτέ να γνωρίζουν ότι οι ε, ε, Ευρωπαίοι αγρότε ε, παράγουν προϊόντα με τον πιο ποιοτικό τρόπο και ακολουθώντας πολύ αυστηρά και ποιοτικά κριτήρια. Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες παρερμηνίες αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ε, γεωργία και την άπτυξη της υπαίθρου και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιληθούν οι παρεξηγήσεις αυτές αν θέλουμε πραγματικά οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκτιμήσουν περισσότερο την ε, συμβολή των ε, Ευρωπαίων γεωργών, ιδίως στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Περιμένω από τον εισηγητή να γνωρίζω ακόμα περισσότερα πράγματα όσον αφορά το πώς καλύπτονται τα ποιοτικά προϊόντα και πώς μπορεί να προωθηθεί η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής παραγωγής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο σε κάποιες ε, αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην αλυσίδα διανομής, αλλά και σε μια καλύτερη προώθηση των ποιοτικών προϊόντων. Αυτό θα έχει πολύ θετική επίπτωση για τους γεωργού, αλλά θα πρέπει επίσης να καταφέρουμε να πειράσουν περισσότερο θετικά την προώθηση των προϊόντων αυτών σε περισσότερες αγορές. Θα πρέπει επίσης να πούμε προς τους ε, εταίρους μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι διαθέτουμε κάποια πολύ ποιοτικά προϊόντα, καθώ επίση και συγκεκριμένα εξειδικευμένα προϊόντα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τα προϊόντα αυτά τα οποία θα βελτιώσουν, θα προωθήσουν ακόμα περισσότερο το γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε στον, στην ανάπτυξη του οικονομικού τομέα σε πολλά κράτη-μέλη. Στην ε, δική μου, για παράδειγμα, τη χώρα, ορισμένα προϊόντα παρουσίασαν μία αύξηση στις εξαγωγές στις τάξεις του 12%. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει μια πολιτική προώθηση ισχυρή, η οποία θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους καταναλωτές, αλλά και την προώθηση των ίδιων των προϊόντων στην αγορά. Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην πρόθεση ποιοτικών προϊόντων στα σχολεία και ότι θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να φέρουμε πιο κοντά αγρότε και πολίτε. Τέλος, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το πώς ορίζουμε την ποιότητα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιβαρύνουμε περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερα κριτήρια τους γεωργούς. Και θα υποβάλω σχέση με αυτό μια τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Τελευταίος ο ε, Μάρ Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Θα είμαι, ελπίζω και εγώ λακωνική. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα, γιατί δείχνουν τα νούμερα ότι ε, λιγότερο από το 24% των ε, πολιτών γνωρίζουν το λογότυπο της ε, βιολογικής γεωργίας και επίσης το λογότυπο για τις ε, ονομασίες προέλευσης και τις ε, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Πολύ έργο λοιπόν ενημέρωση έχει να γίνει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο για την ποιότητα και την προέλευση. Και εκεί ίσως θα πρέπει τα σχολεία να παίξουν το ρόλο τους να διαπαιδαγωγήσουν του μαθητές, αλλά ίσως ήταν πολλά από τα Θα πρέπει ίσως ε, να σκεφτούμε ότι οι νέοι μπορεί να έχουν πολύ πιο σφαιρική αντίληψη από ότι εμείς που εντοπίζουμε περισσότερο την προσοχή μας στα τοπικά προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι και αν θέλουμε να τους ε, διαπαιδαγωγήσουμε προς τη σωστή μας κατεύθυνση πρώτα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όντως η δική μας κατεύθυνση είναι σωστή. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στο Διευθυντή Πατσέκο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας μας από τον κύριο Μποβέ, τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη, γιατί αυτή τη στιγμή εκπονούμε τις νέες νομοθετικές προτάσεις για το σημείο αυτό, οπότε η έκθεσή σας πραγματικά φτάνει την κατάλληλη στιγμή. Γνωρίζουμε και εμείς την ανάγκη για την καταπροτεραιότητα στήριξη των ποιοτικών προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τα υψηλά, ε, τα υψηλά επίπεδα και τις υψηλές προδιαγραφές των γεωρικών μας προϊόντων. Φυσικά θα πρέπει ταυτόχρονα να αναπτύξουμε και τις αγορές και να ε, βελτιώσουμε την ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των ε, κοινοτικών ε, γεωργικών προϊόντων και εντός και εκτός της κοινοτικής αγοράς, όπως επισήμαναν πολλά μέλη της Επιτροπής σας και συμφωνούμε και εμείς. Επίσης, ενστερνιζόμαστε τη γνώμη του εισηγητού και άλλων μελών της Επιτροπής Γεωργίας, ότι το θέμα των βραχιών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τα μέτρα αυτά και τις βραχές αληθισίδες εφοδιασμού, κυρίως ε, από τα μέτρα της ανάπτυξη πέθρου. Ευχαριστώ και τώρα να ξαναδώσω το λόγο για τις τελικές παρατηρήσεις στον εισηγητή μας, τον κύριο Μποβέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ ε, να πω ότι τώρα έχει ξεκινήσει το έργο και φυσικά περιμένω τις ε, τροπολογίες για να διαβρίνουμε την εμβέλεια της έκθεσης, γιατί όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η έκθεση θα χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που καταρτίζει τις νομοθετικές της προτάσεις. Έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εισακωστούμε από αυτήν. Να κάνω κάποιες ε, διορθώσεις, γιατί φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις για το τι εμπίπτει σε αυτή τη χρηματοδότηση, όταν μιλήσαμε για τις αγορές προϊόντων που αντιμετωπίζουν κρίση. Με αυτή η δημοσιονομική γραμμή προσπάθησε καταρχήν να, ε, διαθέσει τα πλεονάσματα, μετά να ανταποκριθούμε στην υγειονομική κρίση. Τώρα αλλάζουμε. Θα πρέπει η απάντησή μας στην κρίση να μην καλύπτεται, να μην εμπίπτει σε αυτή τη δημοσιονομική γραμμή. Γιατί εδώ είμαστε σε μια θετική διατύπωση. Θέλουμε να προωθήσουμε φυσικά τα ποιοτικά προϊόντα, αλλά με βάση κάποια κριτήρια που θα προσδιορίζονται και σε κοινοτικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Ναι, να υποστηρίξουμε τα προϊόντα που ε, αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά όχι σε αυτό το πλαίσιο. Και ε, το είπαμε αυτό και στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Προσοχή να μην δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των μηνυμάτων ε, για το τι καλύπτει αυτό το νέο σχέδιο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης, το σημείο υπερκμον 8. Έχει έρθει ήδη η συγγήτρια, η Τζούλη Γκίρλιν, και θα αρχίσουμε να μιλάμε για του ε, τους ε, τρόπους υπολογισμού ε, για του ε, λογιστικού κανόνε και σχέδια δράση για τι εκπομπέ και τι απορροφή αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσει γη, τις αλλαγές χρήσεων γη και τη δασοκομεία. Έχουμε λοιπόν ε, την γνωμοδότηση τη κυρία Γκέρλινγκ Αλλαγές λοιπόν ε, χρήση γη ε, και δασοκομεία. Η πρόταση αυτή καθορίζει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο για τον τομέα ε, κυρίως όσον αφορά τι αλλαγέ χρήση γη και τη μελισσοκομεία γιατί αυτά θα μπουν στον περιορισμό του 20% των αερίων του θερμοκηπίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Γκέρλινγκ. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια σχετικά σύντομη έκθεση, η οποία είναι αρκετά σαφής. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να αναλώσουμε πάρα πολύ χρόνο συζητώντας τη. Θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι μολονότι είναι σαφής και άμεση η έκθεση αυτή, είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αν πραγματικά θέλουμε να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα όσον αφορά τι χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γη και τη δασοκομεία, χρειαζόμαστε και ένα καλύτερο σύστημα λογιστική απεικόνηση. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλουμε τα επόμενα χρόνια είναι να μην συμφωνούμε ή να τσακωνόμαστε, αν θέλετε, για τον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζουμε τα αριθμητικά δεδομένα. Θα πρέπει εξ αρχή να καταρτήσουμε και να συμφωνήσουμε μια σωστή μεθοδολογία, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστα νούμερα στο μέλλον. Είμαι λοιπόν σαφώς υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι η πρόταση είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, κινείται πάνω στη σωστή κατεύθυνση. Έκανα μία σειρά αλλαγών, την οποία θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω. Ο πρώτος σημαντικός τομέας έχει να κάνει με τα εθνικά σχέδια δράσης, άρθρα, άρθρο 10 και παράρτημα 4 αποφάσισα στη γνωμοδότηση να διαγράψω τα εθνικά σχέδια δράση, γιατί θεωρώ ότι υπερβαίνουν τον αρχικό στόχο. Αν παραμείνουν στο κείμενο, θα πρέπει να είναι καθαρά θελοντικά και πολύ πιο ευέλικτα στη φύση του. Νομίζω το χρονικό περιθώριο των έξι μηνών προβλέπει για τα εθνικά σχέδια δράση είναι ιδιαίτερα στενό για τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα γραφειοκρατικό το ολοπλαίσιο ανταπόκριση στι απαιτήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ουσιαστικά θα ενθαρρύνει πολλά κράτη-μέλη να μην εφαρμόσουν το σύστημα αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή δεν θα συμφωνήσει με την άποψή μου αυτή. Μπορώ να συμβαστώ πάντως σε αυτό το σημείο κίνησής μου όσον αφορά την δική μου τοποθέτηση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η γνωμοδότηση είναι το ζήτημα της ευθυγράμμισης του LULUCF με τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως με την συμφωνία του Ντέρμπαν. Ξέρω ότι η πρόταση αυτή γράφει πριν την τελευταία συμφωνία COP17. Προσπάθησα λοιπόν μέσα στο κείμενο αυτό να ευθυγραμμιστώ με την σύμβαση αυτή του Ντέρμπαν. Αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με κάποιες αλλαγές στα άρθρα 2 ορισμοί και στο άρθρο 9 όσον αφορά τους κανόνες λογιστικής απεικόνησης και έχουμε έπειτα τι κατεξοδότηση πράξης. Γνωρίζω ότι το ζήτημα των κατεξοδότηση πράξεων είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και έχει οδηγήσει πολλές φορές σε αντιπαράθεση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να κάνω κάποιες προσαρμογές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο άρθρο 4 έχω προτείνει κάποιες διαγραφές στους γενικούς λογιστικούς κανόνες ή στους διαχειριστικούς κανόνες λογιστικής απεικόνησης. Σε άλλες περιπτώσεις, έχω, όπως το άρθρο 9.5, έχω προσπαθήσει να παρακάμψω την απέτηση που προβλέπεται, χρησιμοποιώντας τη φράση «minor changes». Και αυτό γιατί πιστεύω ότι οι, οι αλλαγές αυτές είναι πολιτικής φύσης. Επομένως, οι συνομοθέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθούν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για τις αλλαγές αυτές. Και ολοκληρώνω τις παρατηρήσεις στο σημείο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο κυρία Γκέρλινγκ και τώρα λοιπόν α, τη συζήτηση. Αρκετοί έχουν ζητήσει το λόγο. Ειδικά οι συντονιστέ να μην μιλήσουν πολύ για να κάνουμε μετά τι συνεδρίε των συντονιστών. Κυρία Πόλσεν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ντουρμπανοποίηση, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, αυτή τη συζήτηση για την ευθυγράμμιση με τη σύμβαση του Ντέρμπαν. είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση αυτή. Έχω μία μόνο παρατήρηση. Στην Ευρώπη, όταν μιλούμε για δασοκομεία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών για τον κλάδο αυτό. Άλλα προβλήματα έχουμε τα δάση οι νότιες χώρες και άλλα προβλήματα έχουμε τη δασοκομεία οι βόρειες χώρες. Στην Νότια Ευρώπη ε, φυτεύουν όλο και περισσότερα δάση προσπαθώντας να διατηρήσουν ε, τα δάση που υπάρχουν ε, και που απειλούνται από την ανοβρία, τη μεγάλη ξηρασία και τις πυρκαγιές που μαστίζουν τα δάση στις νότιες χώρες. Στην Βαλένσια, για παράδειγμα, έχουμε αυτόν τον καιρό πολύ εκτεταμένες πυρκαγιές, δυστυχώς, και δημιουργείται ένα τεράστιο κλιματικό πρόβλημα. Και είναι σημαντικό φυσικά να κατασβεστούν αυτές οι πυρκαγιές, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά επαναλαμβάνω, ε, κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετική κατάσταση. Στη δική μου πατρίδα έχουμε τελείως διαφορετικά προβλήματα ως προς τη δασοκομεία. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, αποθήκευση, τη δέσμευση και αποθήκευση του άθρακα. Γιατί εμείς έχουμε η υπερβολική ήγρανση των ε, δασών. Έχουμε, έχουμε αντίθετο <laughs> πρόβλημα δηλαδή από αυτό τις ξηρασίες που αντιμετωπίζει ο Νότος. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κοινού κανόνε. Έχετε όμω υπόψη ότι αυτοί οι κοινοί κανόνε θα ισχύσουν για πολύ διαφορετικέ πραγματικότητε. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τοπική και περιφερειακή διάσταση σε αυτή τη λογιστική απεικόνηση, σε αυτού του λογιστικού κανόνε. Ευχαριστούμε, κυρία Πόλσεν. Ε, κυρία Κέστιγκερ και μετά ο Άγνιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγητρία για την πολύ καλή δουλειά τη. και την προσέγγιση τη δική της την έκθεση την βρίσκω πάρα πολύ καλή. Η στόχη, κατά την άποψή μου είναι αδιαμφισβήτητοι με το Λουλουτσεεφ αλλά όπως ε, πολύ συχνά ακούμε το να έχει κανείς ε, καλές προθέσεις δεν αρκεί. Ε, χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που η συγγήτρια επισημαίνει ότι πρέπει να είναι σωστή η αριθμή αυτό το προτινόμενο σύστημα δικτών, κατά την άποψή μου, πρέπει να τύχει επεξεργασίας, διότι επουδενή ε, δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη να έχουμε πολλά και διαφορετικά συστήματα στη δασοκομεία. Γιατί η δασοκομεία ε, προσφέρει ένα τεράστιο δυναμικό για την παραγωγή βιομάζας. Ε, δεν είναι δηλαδή δυνατόν να υπάρχουν και προγράμματα όπου παραγωνίζεται πλήρως η δασοκομεία. Θέλω να επισημάνω ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει επουδενή να συμβεί. Έχω ουσιαστικές επιφυλάξεις όσον αφορά τη γραφειοκρατία η οποία ε, προκύπτει από αυτό το σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, επισημάνω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν και οι διαπραγματεύσεις ε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν τη γεωργία και νομίζω ότι ε, ρόλο παίζει και η σχέση κόστους κόστους-οφέλους. Αυτά που είπε η συγγήτρια για τα εθνικά προγράμματα δράσης τα υπογραμμίζω ανεπιφύλακτα. Εγώ είμαι ε, αμύντορας αυτών των ε, συστημάτων ε, και όσον αφορά την παραγωγή μας, ας μην ξεχνάμε ότι το σημαντικότερο από όλα είναι να υπάρχουν κίνητρα. Εγώ ε, στηρίζω ανεπιφύλακτα τα κίνητρα. Στον τομέα της γεωργίας νομίζω ότι με τα κίνητρα θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από το να εξαναγκάζουμε τους γεωργούς ε, και όσοι ασχολούνται με τα σοκομεία να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει στις αρμοδίες των κρατών μελών και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει ένα στρογγύλεμα όλης αυτής της κατάστασης. Ευχαριστούμε πολύ. Αγνιού και πάλι Μακίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι από μένα περιμένετε κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Ο τίτλος και μόνο ο τίτλος αρκεί για να κάνει οποιοδήποτε αγρότη να ανατριχιάσει. Λέει «Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράση για τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης». Εδώ η γραφειοκρατία αποκτά ένα νέο όνομα. Ο Γεωργός θα πρέπει να υπολογίσει πόσο εκπέμπει τα ζώα του και να τα περιορίσει. Τι γίνεται με την... Ε, εντάξει, με την εντατική κτηνοτροφία που γίνεται στο εσωτερικό το καταλάβω, αλλά με την εκτατική κτηνοτροφία στην Ήπεθρο πώς θα τα υπολογίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους δυσκολεύουμε όλο και περισσότερο τη ζωή. Μεθάνιο περισσότερο εκπέμπεται από τα παρθένα δάση, τα τροπικά δράση που όμως ε, το ε, πράσινο λόμπι προσπαθεί να προστατεύσει. Νομίζω ότι είναι γελία αυτή η πρόταση. Οτιδήποτε ε, παράγεται σε μια καλλιέργεια απορροφά αέρια του θερμοκηπίου και άρα θα έχουμε και πιο γρήγορη βλάστηση. Επίσης, έχουμε υψηλά επίπεδα διοξίδιου του άνθρακα αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα σχέση με 30 χρόνια. και Παρόλα αυτά, παρόλο που έχουμε όμως ε, ε, ε, οι ειδικοί πρόβλεψαν ε, ζεστά καλοκαίρια και κρύους χειμώνες, ε, τι να πω, δεν έχουμε αυτά που μας περίμεναν. Ε, βλέπω ότι έχουμε πολύ περισσότερο από το μέσο όρο των βροχοπτώσεων και τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο και Φαίνεται ότι είναι τελείως παράλογες αυτές οι θεωρίες στο Γεωργικό Υπουργείο της ΔΕΦΡΑ που πραγματικά έχουν διαψευστεί παταγωδός. Έχουμε αποτύχει να... Βέβαια το θέμα της αποτυχίας της καταμέτρησης του μεθανίου των κοπαδιών μου θα θεωρηθεί ως σφάλμα και ως έλλειψη συμμόρφωσης. Ίσως θα πρέπει να επενδύσω σε, μια συσκευή, ε, ε, σε ένα μετρητή της μυρωδιάς, ένα μυρωδομετρητή. Ίσως αυτό θα πρέπει να κάνω. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκάρλινγκ για την πολύ καλή παρουσίαση και για την έκθεσή της. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς μετά όσα είπε ο κύριος Άγνιος όσον αφορά την αντίδραση των αγροτών. Ουσιαστικά και η δική μου άποψη ομοιάζει με αυτή του κυρίου Άγνιου στην πράξη πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία προτείνονται εδώ πέρα. Και όσοι δεν έχουν διαβάσει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας παρακαλώ πολύ να το κάνουν, γιατί πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ την εργασία των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί ότι είναι πολύ θετικό να γίνουν οι αλλαγές αυτές, πάντως πιστεύω ότι θα οδηγήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο γραφειοκρατίας για τους γεωργούς. Συμφωνώ με την προσέγγιση της κυρίας Γκάρλινγκ ότι πολλές φορές τα όσα προ, προβλέπονται για τα εθνικά σχέδια δράσης είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικά. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση όμως να καταγράψουμε σωστά την γεωργική δραστηριότητα και αυτή η υποχρεωτική επιβολή εκθέσεων όσον αφορά τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για το 2013 θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να μελετήσουν πολύ προσεκτικά την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα τη συζητήσουμε αργότερα σήμερα το βράδυ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή και από την δική σας την Επιτροπή. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη συντάκτρια της εκδομοδότησης για την προσοχή που ήδη έδωσε και εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες προκειμένου να γίνει μια πολύ σημαντική συζήτηση για το ζήτημα αυτό, για την έκθεση αυτή και να μην περάσει έτσι χωρίς έλεγχο και χωρίς τροπολογίες. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που έλεγξαν. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά την πρόταση τη Επιτροπή. Και με αυτή την ευκαιρία θα δώσουμε αμέσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, που είναι ο κύριος Χόλσεν από την ε, Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, όχι περιβάλλοντος, κλίματος, Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για την ε, πολύ αξιέπαινη της προσπάθεια. Όντως δεν είναι και πολύ προσιτό αυτό το θέμα. Υπάρχει πολλά, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα, υπάρχουν πολλές ακρονιμίες που προέκυψαν από διεθνείς διαπραγματεύσεις. Άκρος τεχνικό το ζήτημα, αλλά η εισηγήτρια πραγματικά κατάφερε να συμπεριλάβει και τέτοιες συντομεύσεις τεχνικές με πολύ αξιέπαινο τρόπο. Αναφέρθηκε ντορμπανοποίηση της έκθεσης και ευχαριστώ για την προσπάθεια αυτή με τη συμφωνία του Ντέρμπαν που έκανε η συγκήτρια. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πρόταση αυτή αφορά μία απόφαση για τους λογιστικούς κανόνες. Δηλαδή θα ισχύσει μόνο για τους αξιωματούχους των κρατών μελών, για τα, για συστήματα των κρατών μελών. Πρόκειται για λογιστικούς κανόνες που στην πράξη ε, αφορά το πώς ε, λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα στοιχεία τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά μέτρα εδώ, ούτε θα επιβληθούν γραφειοκρατικές απαιτήσει ε, στους γεωργούς. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αφορά μόνο τα συστήματα, τα λογιστικά των κρατών μελών. Και ουσιαστικά εφηγραμμιζόμαστε με τη συμφωνία του Ντέρμαν για το πώς θα ομαδοποιηθούν κάποια στοιχεία σε ένα, σε ένα κυβερνητικό σύστημα λογιστικό. Περί αυτού μόνο πρόκειται. Πάντως ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Περιμένουμε και τη συνέχεια των συζητήσεων και γενικώ σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, για το κλίμα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την Julie Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε, όντως υπάρχουν κάποια ζητήματα για τη δασοκομεία. Γι' αυτά προφανώς μπορείτε να στείλετε τροπολογίες και να συζητήσουμε περισσότερο τα όσα είπατε. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν. Να ευχαριστήσω επίση όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Πέρα από τον κύριο Άγνιου βέβαια, αλλά ποτέ δεν είναι καλός μαζί μου, ούτως ή άλλως. Θα ήθελα να πω ότι η Γενική Διεύθυνση Κλιματικών Αλλαγών μας είπε ότι δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε εξατομικευμένες γεωργικές εκμετέλευσεις, αλλά αναφερόμαστε ουσιαστικά στα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη στον λογιστικό έλεγχο των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω τις ανησυχίε τη κυρία Μαγκίνες και του κυρίου Άγνιου ότι αν τελικά όλα πάνε κατευχήν, ενδεχομένως να επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση η Κλίμα μπορεί στο μέλλον να καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή τα οποία τροποποιούνται στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι ευθύνη μου στα πλαίσια της Επιτροπής Γεωργίας είναι να παραμείνει το κείμενο αυτό ως το δυνατόν πιο απλό πιο άμεσο. Παρακολούθησε επίσης τις συζητήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και είδα εκεί πέρα ότι το κείμενο θέλουν να το κάνουν πιο πολύπλοκο, πιο δύσκολο και πολλές φορές ε, πιο άκαμπτο. Η έκθεση μου λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ άμεση και απλή και αναφίβολα θα συζητήσουμε και πάλι στο μέλλον την έκθεση αυτή αφού ξεπεράσουμε πρώτα τις βασικές δυσκολίες που έχουν προκύψει με τις μεθόδους λογιστικής. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Για λίγο έχει ζητήσει το λόγο ο Άλμπερτ και έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση προς την εισηγήτρια. Μόλις διάβασα ότι παλαιότερα στη Βόρεια Αμερική υπήρχαν 200 εκατομμύρια βίζονες ε, ε, οι οποίοι είχαν τεράστιες ε, ποσότητες εκπομπών μεθανίου. Το 1900 υπήρχαν μόνο 300 βίζονες και γιατί τους εξαφάνισαν, μήπως με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν στην αλλαγή του κλίματος και στις αλλαγέ που υπήρξαν γενικότερα. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε, Τζουλ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχει κλείσει το όλο θέμα. 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ε, είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση απολογιών για την έκθεση Γκέρλινγκ και θέλω να σας πω ότι όσον αφορά στην ε, έκθεση Μποβέ, η τροπολογία, η καταληπτική ημερομηνία είναι 29 Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε όλους και τώρα λοιπόν λύεται η συλλεντρίαση και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.30. 9.30. Και τώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Grazie.